Good. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Λοιπόν, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε. Πριν ε, ξεκινήσουν οι εργασίες μας, ε, οι διερμηνείς θέλουν να σας πω κάποια πράγματα. Όπως έχετε ίσως ακούσει, βρισκόμαστε στην 35η ε, μέρα κινητοποιήσεων και άρα μέχρι να λυθεί η εργασιακή διαμάχη, έτσι και σήμερα η συνεδρία θα τελειώσει ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα χωρί υπέρβαση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια γνωρίζουμε την κατάσταση και ελπίζουμε η διοίκηση να βρει μια λύση προσεχώ. Λοιπόν, πρώτο θέμα, έγκριση τη ημερήσια διάταξη Υπάρχουν ετοίματα για να αλλάξει, όχι, οπότε εγκρίνεται χωρί αλλαγέ. Σημείο 2. Τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 20-21ης Ιουνίου 2018. Εάν ε, δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης, τα πρακτικά εγκρίνονται. Σημείο 3. Η απόφαση, η απόφαση των συντονιστών. Στι 20 Ιουνίου. Η ίδια διαδικασία ισχύει και εδώ, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει ε, εγκρίνονται. Μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Και σημείο 4. Ω συνήθω η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους επισκέπτες μας ε, από την Λιζαφόνα μέχρι το Λούνεμπουργκ και από το Ελσίνκι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε διερμηνία. Οπότε... Παρακαλώ να μιλάτε δυνατά, καθαρά και αργά για να σας ακούν όλοι. Και ερχόμαστε έτσι στο σημείο 5. Το βασικό θέμα της σημερινής ημέρας η δημόσια ακρόαση μας για την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια συμφωνία εταιρική σχέσης. θα θέλαμε να δούμε πιο προσεκτικά αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώς ο Ζαν Λουκ δεν είναι εδώ. καταφθάνει. Μου λένε... Όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε την εμπορική συμφωνία και τις πρόπτικες της συμφωνίας και αρχικά ε, πρέπει να ε, έχει υπογραφεί 11 Ιουλίου λόγω όμω των πλημμυρών στην Ιαπωνία αναβλήθηκε και θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα της πλημμύρας Thanks a lot. Σας ευχαριστώ. Είναι λοιπόν σαφές πως εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας προς τους οικείους των θυμάτων. Την Παρασκευή που μας πέρασε το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως ε, για την υπογραφή. Οπότε από την ευρωπαϊκή πλευρά όλα είναι έτοιμα για να υπογράψουμε την συμφωνία και να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προς ακύρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι το τελευταίο αλλά το σημαντικότερο θεσμικό όργανο της όλης ε, διαδικασίας. Εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Και βεβαίω η σημερινή ακρόαση είναι ένα πρώτο βήμα στην ανάπτυξη των συστάσεων των δικών μας για την συμφωνία και βεβαίως θα έχουμε κάποιο ψήφισμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, συνένεσης ε, για να επισημάνουμε και την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κύρωση αυτή. Οπότε τους επόμενους μήνες θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και χωρίς ε, βιασύνη την συμφωνία αυτή και άρα Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Αλλά πρόκειται για την αρχή και όχι το τέλος της διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, αναλόγως με το πώς θα προχωρήσουμε. Η Επιτροπή μας έχει ε, εμπλακεί στο θέμα αυτό. στην θέση που είχε λάβει το Κοινοβούλιο το 2012 κάναμε δύο αντιπροσωπείες ε, το 2011-2015 στην Ιαπωνία και θα ξαναταξιδέψουμε τον Σεπτέμβριο φέτος είχαμε πολλές ε, συζητήσεις με το Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Εμπορίου και με την Επίτροπο την ίδια έγινε ένα εργαστήριο που οργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής και πολλές μελέτες για το θέμα αυτό. Και βεβαίως, το σημαντικότερη δουλειά επί του θέματος, είναι στην ομάδα παρακολούθησης υπό την Προεδρία του μόνιμου εισηγητή του κυρίου Σίλβα Περέιρα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η ομάδα αυτή συνεδρίασε 21 φορές εάν δεν κάνω λάθος. δηλαδή για πραγματική, πραγματικά στενή παρακολούθηση και επιρροή της διαδικασίας οπωσδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως επειδή εργαζόμαστε με διαφάνεια η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου όπως και το κείμενο άλλωστε της συμφωνίας και είχαμε πολλές επαφές με πολλούς ενδιαφερόμενους όσον αφορά την συμφωνία και το κείμενο που έχουμε τώρα επιτάπητος κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο ζητήματα που εκκρεμούν το ένα είναι βεβαίως το ζήτημα της κύρωσης των δύο συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας η 111 για την καταναγκαστική εργασία και 105 για την της διακρίσης του ε, και υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης για τις ροές ε, δεδομένων που λέει ότι μετά από τρία χρόνια μετά την θέση ενισχύ της ε, συμφωνίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή. Αυτά λοιπόν φαντάζομαι θα συζητηθούν. το πρώτο θέμα. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Ζαν Λουκ Ντεμαρτή, Γενικό Διευθυντή Εμπορίου και τον κύριο Σουζούκη, Ειδικό Συμβουλό του Υπουργείου των Εξωτερικών και πρώην επικεφαλής διαπραγματευτή της Ιαπωνίας για την συμφωνία αυτήν. Καλώς ήρθατε. Πριν δώσω τον λόγο στον Ζαν θα ήθελα να ζητήσω από τον μόνιμο εισηγητή, τον ε, κύριο Σίλβα Περίερα, να μας κάνει μια εισαγωγή. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν, επιτρέψατε μου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τις αρχές της Ιαπωνίας και τους πολίτες που υπήρξαν θύματα των πρόσφατων πλημμυρών στην ε, δυτική περιοχή της Ιαπωνίας ήταν μεγάλο πλήγμα και ελπίζουμε οι επιχειρήσεις διάσωσης να είναι πετυχημένες. Όσον αφορά τη σημερινή ημερήσια διάταξη, επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ήρθαν εδώ, ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας που έκαναν το μακρύ ταξίδι από την Ιαπωνία για να μας εκφράσουν τις απόψεις για την εμπορική συμφωνία, τον κύριο Σουτζούκη, τον κύριο Σιμίζο και τον κύριο Καβασίμα. Ιδιαίτερε ευχαριστίες στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας που διοργάνωσε τα πάντα ούτω ώστε να μπορέσει να παραστεί εδώ ο κύριο ε, Σουτζούκι. Και ε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην Ιαπωνική κυβέρνηση. Και καλώς ήρθατε προς όλους. Όπως γνωρίζετε, ε, στην, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία λέξη όσον αφορά την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας και θεωρούμε τη δημόσια αυτή ακρόαση ότι έρχεται σε κατάλληλη στιγμή και είναι ιδιαίτερο σημαντική. Γιατί στι 6 Ιουλίου το Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να υπογράψει τη συμφωνία και ε, αλλά θα πρέπει να θεσπιστεί μια νέα ημερομηνία για την υπογραφή. Ε, Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία επιθυμούν ε, το συντομότερο δυνατό να υπογραφεί η συμφωνία αυτή και αυτό σημαίνει ότι για το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση τους προσεχείς μήνες σχέση με το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως παίρνει πολύ σοβαρά αυτό το έργο και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το έργο του Κοινοβουλίου δεν ξεκίνησε με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αλλά πολύ νωρίτερα στη διαδικασία ε, και έγινε ένα ψήφισμα ε, τον Οκτώβριο, εκπονήθηκε όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή και όπως ξέρετε συστάθηκαν και πολλές ε, επιτροπές ε, παρακολούθησης της Διεθνούς Επιτροπής ε, Εμπορίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δύο βασικά έργα να οριστικοποιήσει το τελικό κείμενο της, σύμφωνη, της συμφωνίας και να ακούσει όλους τους, να διαβοληθεί με τους ενεχόμενους φορείς. Ε, το έργο αυτό ξεκίνησε ήδη στην ομάδα παρακολούθησης ε, και στην ίντα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να λεφθεί αυτή η συζήτηση. Η εντολή έχει δημοσιευθεί. Το ε, και η συμφωνία αυτή πραγματικά αξίζει να συζητηθεί εις βάθος. Θα ήθελα να αναφέρω στην το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται σε αυτή τη φάση μετά τη συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, τον Αύγουστο το σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο σύστασης θα ε, υπάρχει το Δεκέμβριο Έχουμε μία αποστολή ε, στην Ιαπωνία το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα εξετάσουμε το σχέδιο σύστασης τέλη Σεπτεμβρίου και προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 2 Οκτωβρίου και επίσης για να έχουμε την γνωμοδότηση των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών η ημερομηνία είναι 11 Οκτωβρίου. Βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, μπορεί να διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου και η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Σήμερα έχουμε λοιπόν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε τους διαπραγματευτές και Επίση, του διάφορου ενδεχόμενου ε, φορεί και ενδιαφερόμενους για την εμπορική συμφωνία και θα ακούσουμε ιδιαίτερω τι σημαίνει για τους εμπορικούς ε, κύκλου αλλά και για τους πολίτε. Τέσσερα βασικά θέματα αναμένεται να συζητηθούν εδώ. Βεβαίω η διάσταση στρατηγική, η στρατηγική διάσταση της συμφωνίας σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων του διεθνούς που αντιμετωπίζει το Διεθνέ εμπόριο η οικονομική πτυχή βεβαίως της συμφωνίας, γιατί ε, πάντοτε ε, ενδιαφέρει τις αξιολογήσεις και ε, το γεγονός ότι το εμπόριο ενέχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών και θα πρέπει να τηρούνται βεβαίως οι προδιαγραφές ε, των συμβάσεων του ILO για τις εντρικές εργασίες και θα συζητηθεί βεβαίως ε, το ζήτημα των, ε, τι θα πρέπει να αναμένουμε από την Ιαπωνική κυβέρνηση όσον αφορά την επικύρωση αυτών των συμβάσεων. Ε, θα... Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο για 10 λεπτά στον Ζαν Λουκ να μας κάνει μια εισαγωγή. Thank you very much, uh, Bernd. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, και πραγματικά είναι μια εποχή εξαιρετικά παράδοξη, γιατί ποτέ οι πολίτες δεν έχουν υποφεληθεί τόσο πολύ από το εμπόριο και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί τόσο πολύ ένα αφιβόλο η πολιτική εμπορίου. Ε, ε, και βεβαίως υπάρχουν πολλές σημαντικές ε, απειλές και υπονομεύεται το πολυμερές σύστημα εμπορίου. Και περάσαμε το πρώτο ήμιση της εντολής της Επιτροπής, προσπαθώντας να βάλουμε σε τάξη του Κοινοβουλίου, γιατί έγιναν ε, κριτικές όσον αφορά την ε, πολιτική εμπορίου. Ορισμένοι κατηγόρησαν την πολιτική εμπορίου να είναι υπερβολικά, ότι είναι υπερβολικά αδιαφανής. Ε, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με τη λήψη μέτρων όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ορισμένοι είπαν ότι επικεντρώνεται υπερβολικά η πολιτική μας στο οικονομικό κέρδος. Τώρα έχουμε κάποια κεφάλαια ε, στις, ε, στην πολιτική μας, οι οποίες ε, θα προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Και πέρα από αυτό προσπαθούμε να επιλύσουμε όλα τα θέματα που εκκρεμούν. Υπάρχει σαφήνως αναφορά της τις αλλά και της εθνικές αρμοδιότητες βάσει του Δικαστηρίου της Σιγκαπούρης. Ε, και προωθούμε τις πιο σύγχρονες ε, τεχνολογίες καθώς και, και εκπονούμε μηχανισμούς επονδύσεων ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις τρευλώσεις του εμπορίου με σύγχρονα εργαλεία προάσπισης ε, των μηχανισμών εμπορίου. Προσπαθούμε να εξάσουμε προσοχή τις σύγχρονες προκλήσεις και αυτό μας καθιστά έναν προβλέψιμο εταίρο ο οποίος μπορεί αποτελεσματικά να εκπληρώσει τα, τα να ακολουθήσει τα συμφέροντά του. Ε, τώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ιαπωνία γιατί πρόσφατα έγιναν ε, πλημμύρες, ε, υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και πολλά θύματα και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας προς τις ε, Ιαπωνικές αρχές και τους πολίτες της Ιαπωνίας. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και ο Πρωθυπουργό ΑΠΕ έλαβε μέτρα κατεπίγουσας ε, ανάγκης. Ε, εμείς ε, βρισκόμαστε στο πλευρό των Ιαπώνων ε, συμμάχων μας που υπήρξαν θύματα αυτής της φυσικής καταστραφής. Ο Πρωθυπουργός Ιαπωνίας, ο κύριος Ιούνκερ και ο, και κύριος Τάσκα ε, αποφάσισαν ότι η συνάντηση για την υπογραφή της συμφωνίας θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα στο, στο Τόκιο. και αντανακλά ακριβώς την ε, σημασία της συμφωνίας αυτής τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ιαπωνία. Η Επιτροπή θέλει να ε, επισπεύσει την ε, διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας ούτως ώστε να μπορέσουν να ευεργετηθούν και τα δύο μέρη. Και αυτό θα πρέπει να μας εκπλήσει γιατί είναι η Ιαπωνία ο δεύτερος πιο σημαντικός εμπορικός μας εταίρος μετά την Κίνα στην Ασία. Και πάντα και πριν από αυτή τη συμφωνία η Ιαπωνία ε, ήταν εξαιρετικά σημαντική και πρόκειται για μια ε, πολύ σημαντική, μεγάλη εμπορική ε, συμφωνία, η πιο σημαντική που έχει υπογραφεί και εφόσον επικυρωθεί θα καλύπτει ένα τρίτο του παγκοσμίου ΑΕΠ. Και όταν η συμφωνία αυτή προσλάβει το πλήρες της ε, δυναμικό, ε, το 94% των ιαπωνικών εισαγωγών θα είναι απολύτως ε, ελεύθερο. Η Ιαπωνία έχει μια προστατευμένη αγορά, 50% στα κρασιά, 40% στο τυρί, στις σοκολάτες κλπ. Ε, η συμφωνία λοιπόν θα είναι εξαιρετικά σημαντική εδώ. Ε, τα, η αυτοκινητοβιομηχανία θα απελευθερωθεί σε μια μεταβατική περίοδο 7 ετών. Η συμφωνία αυτή με την Ιαπωνία δείχνει ότι προσπαθούμε να ξεχρονίσουμε την εμπορική μας ε, πολιτική και πραγματικά διανοίγει και νέους ε, τομείς. Όσον αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες, ε, εξασφαλίζουμε μία ρήτρα ασφαλείας για, τις, για τους ιαπωνικούς σιδηροδρόμους και μετά από αυτό θα διευρυνθεί σε 7 πόλεις το σιδηρονομικό δίκτυο της Ιαπωνίας. Γιατί για πολλά χρόνια διαφορετικές προδιαγραφές της Ιαπωνίας είχαν παρεμποδίσει τις εξαγωγές μας. Τώρα ε, ελπίζουμε η συμφωνία αυτή να είναι υποδηματική όσον αφορά το άνοιγμα ε, των αγορών. Ε, θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε τομείς κλειδί όπως είναι ο τομέας ο φοπλιστικός κλπ. Ε, τον πλοίων, συγγνώμη. Μια δεύτερη συνάντηση με τον βασικό διαπραγματευτή θα λάβει χώρα εδώ στις Βρυξέλλες και είναι σημαντικό ότι, και επιμένουμε σε αυτό ότι δεν θα υπάρξει καμία πιστοδρόμηση προς ε, το παλαιό καθεστώς. Η συμφωνία αυτή επίσης σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα, τις γεωγραφικές ε, ενδείξεις ε, προέλευσης και υπάρχει προστασία για πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι τοπικές ενδείξεις θα, θα έχουν πλήρη ε, προστασία. Και ε, το θέμα της εταιρική ε, διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία αυτή και υπάρχουν και άλλα κεφάλαια τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί η Ιαπωνία είναι εντελώς διαφορετική αγορά από τη δική μας η γλώσσα ε, και τα ήθη και οι εμπορικές ε, συνήθειες αποτελούν πρόκληση για τους Ευρωπαίους και οι ελληνικοί δασμοί καθιστούν ε, το βίο για μας ακόμα δυσχερέστερο. Ωστόσο, τα κεφάλαια αυτά μας δεσμεύουν να ενημερώσουμε πλήρως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και έχουμε φτιάξει σημεία επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και αυτά αφορά και τους ε, καπνοπαραγωγούς, αλλά βεβαίως όλα αυτά χρειάζουν περαιτέρω βελτιώσεων. αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία της συμφωνίας μας. Μπορούσα να περάσω όλη τη μέρα στην συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς διμερής, αλλά αποστάλει ένα, παγκόσμιο, ένα μήνυμα παγκοσμίω. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συναντιούνται υπέρ της παγκοσμιοποίησης, του ανοιχτού εμπορίου και προκειμένου να εγκρίνουν κανόνες που να είναι θεμητοί για όλους. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτές τις ε, μέρες όπου υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ε, για το διεθνές σύστημα εμπορίου το οποίο ε, έχει ανθίσει εδώ και πολλά χρόνια. Ε, η μεγαλύτερη απειλή βεβαίω προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε και είναι ανάγκη η Ιαπωνία να συμμαχίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να, που σχετίζονται με τις ΗΠΑ θα πρέπει να παρασυγγιστούν βάσει των ρυθμίσεων και των κανόνων του ΠΟΕ. Ε, έστω και αν ορισμένοι θέλουν να αποχωρήσουν από το Διεθνές Σύστημα Εμπορίου, ωστόσο η Επωνία ε, τίθεται στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μάχη κατά του προστατευτισμού. Τα στρατηγικά και τα οικονομικά ωφέλη αυτής της συμφωνίας είναι απολύτως ξεκάθαρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Περέιρα, την εισηγήτρια, καθώς και την Επιτροπή Ίντα για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις, γιατί ε, η σφορά τους ήταν ε, πολύτιμη. Ε, στις διαπραγματεύσεις. Ε, σημαντικές ε, πληροφορίες μας δόθηκαν από την Επιτροπή αυτή σε σχέση με την Ιωπωνία και η συνεργασία αυτή επικυρώνει την προσήλωση στις αρχές της Συμφωνίας των Παρισίων. Και είναι η πρώτη συμφωνία αυτή με την Ιαπωνία η οποία θα συνάπτεται μετά τη σύναψη της ε, Συμφωνίας των Παρισίων. Ελπίζουμε λοιπόν να επικριθεί πολύ σύντομα ε, και η ψηφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιτρέψει την ε, ταχεία θέση ισχύ αυτής της συμφωνίας. Η αποστολή του Κοινοβουλίου στην Ιαπωνία επίσης θα είναι σημαντική. Ελπίζω να συνδεθείτε με όλους τους σημαντικούς, μας, ε, σημαντικούς εταίρους ε, στην Ιαπωνία. Και θα ήθελα την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω τον πρέσβη κύριο Σουτζούκη, ο οποίος είναι παρόν εδώ καθώς ε, και το Γενικό Διευθυντή της, ε, ε, για το κλίμα, της Γενικής Διεύθυνσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συμμετείχε επίσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σκοπιά της ευρωπαϊκής πλευράς και θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Σουζούκη για να μας πει τα της ιαπωνικής πλευράς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σίλβα Περέιρα, Μονή εισηγητή για την Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα εξ ονόματος της κυβέρνησης και του Ιαπωνικού λαού να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ελληνική την οποία εκφράσατε εδώ σήμερα για όσους υπέφεραν από τις πρόσφατες ε, δυνατές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία. Η πρόβλεψη οπωσδήποτε μας έλεγε ότι θα έχουμε ε, δυνατές βροχοπτώσεις που δεν είχαν ξαναεμφανιστεί αλλά ε, ξεπέρασε και τις προβλέψεις τελικά η βροχοπτώση. Δυστυχώς είχαμε πολλά θύματα οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αισθήματα αυτά αλληλεγγύης και ελπίζω να μπορέσουμε να ανακάμψουμε το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπε και ο κύριος Ντεμαρτή, η υπογραφή της ε, συμφωνίας αναβλήθηκε, αλλά όχι πολύ, θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα και από την δική μας την πλευρά επίσης ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στείλουμε το κείμενο αμέσω ε, στο Κοινοβουλίο για τις δικές τους διαβουλεύσεις. Πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν από τον κύριο Ντεμαρτή και στην δική μας ε, την διαπραγμάτευση της οποίας ηγήθηκα τους τελευταίους 12 μήνες η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάλυψαν πως έχουμε πάρα πολλά κοινά οπότε πολλά από τα σημεία αυτά ήδη αναφέρθηκαν ε, θα προσπαθήσω να επαναλάβω αρκετά από αυτά αλλά θα ήθελα να πω ε, ευθύς εξ αρχής ότι όπως αναφέρθηκε για εμάς η σημασία αυτής της ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης πηγαίνει πολύ πιο πέρα από το ελεύθερο εμπόριο. Είναι ένα μέσο ώστε η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουν ένα ανοιχτό οικονομικό σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε δίκαιους και ισορροπημένους κανόνες. Και αυτό είναι ε, όλο και σημαντικότερο καθώς βλέπουμε μια κάποια σύγχυση θα έλεγα στον κόσμο του εμπορίου ταυτόχρονα μαζί με την Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που θα υπογραφεί την ίδια στιγμή είναι ένα σημαντικό μέσο για να ενισχύσουμε την σχέση μας την στρατηγική μας σχέση είμαστε ενωμένοι ε, αυτήν την κοινή έννοια σεβασμού κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα δίκαιο και ανοιχτό οικονομικό σύστημα. Η Ιαπωνία, όπως αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Ντεμάρτη, είχε αναλάβει πολλές ε, πρωτοβουλίες στον τομέα του εμπορίου. Η συμφωνία αυτή είναι μία. Έχουμε άλλες δύο σημαντικές συμφωνίες που προγραμματίζουμε. Μία είναι η συνολική συμφωνία για την διατλαντική την, με την Συμφωνία Εμπορικής Σχέσης του Ειρηνικού και η τρίτη είναι μια περιφερειακή συνολική οικονομική συνεργασία την οποία διαπραγματευόμαστε με 15 άλλους εταίρους στην περιοχή μας ε, της Ασίας και του Ειρηνικού. Και οι τρεις αυτές ε, πρωτοβουλίες καλύπτουν πάνω από το 70% του ιαπωνικού εμπορίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε σύγχυση και χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την περαιτέρω απελευθέρωση η Σύμφωνια εταιρική σχέση, όπως είπε και ο κύριο Ντέμαρτη, καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους και το συνολικό ΑΕΠ είναι περίπου το 1 τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για εμάς για να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία ενός οικονομικού συστήματος ανοιχτού που θα βασίζεται σε κανόνες και θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη ε, ανεπτυγμένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και μιλάμε για δύο προχωρημένες οικονομίες και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα παράδειγμα. Είμαστε σημείο αναφοράς για άλλες εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική συμφωνία βεβαίω πα... Είναι πάρα πολύ μεγάλη και βεβαίως υπάρχει και η μη δασμολογική πτυχή αυτής της συμφωνίας που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα ωφέλη που σημαίνει η κατάργηση των δασμών. Αλλά να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα άμεσα ωφέλη. Η Ιαπωνία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομική μου και η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη. Οπότε το επίπεδο του εμπορίου δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το οικονομικό μας βάρος. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο 30% των εξαγωγών μας μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά αδασμολόγητες και γύρω στο 7% των ε, ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ο αριθμό αυτός δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Οπότε με τη συμφωνία αυτή αυτό θα αλλάξει. Όπω είπε και ο Σντεμαρτή, μετά από την μεταβατική περίοδο για τα βιομηχανικά προϊόντα 100% των δασμολογικών γραμμών θα είναι δασμολογητές και κάποια προϊόντα και κάποια ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα σε αυτά πάνω από το 95% των δασμολογικών γραμμών θα μηδενιστούν. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους παραγωγούς και εξαγωγείς μας για να ενισχύσουν τις δραστηριότητες τους ε, σε δύο από τις πιο προωθημένες ε, και προχωρημένες αγορές. Δεν θα αυξήσει μόνο τις ευκαιρίες πρόσβασης ε, στην αγορά, θα δημιουργήσει και ευκαιρίες, παραδείγματο χάρη στην ανταλλακτικά αυτοκινήτων για τις ε, αλυσίδες προμηθειών και άρα θα σημαίνει βαθύτερη βιομηχανική συνεργασία. Οπωσδήποτε η Ιαπωνία εξάγει πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως ξέρετε τα και η παραγωγή ευρωπαϊκών ε, ανταλλακτικών είναι σημαντικοί προμηθευτές ε, των Ιαπώνων ε, παραγωγών. Στη Γεωργία επίσης έχει αναφερθεί οπωσδήποτε για το βόλιο, χοιρινό, κρέας, το τυρί, κάποια κατεργασμένα τρόφιμα, ζυμαρικά, σοκολάτα και γλυκά. Θα κερδίσουν πάρα πολλά οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Και στην αρχική φάση, δεν θα αρνηθώ ότι θα ωφεληθούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι παραγωγοί από τους Ιάπωνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσει αυτή η συμφωνία. Η Ιαπωνική Γεωργία αυτή την στιγμή περνάει έναν σημαντικό μετασχηματισμό και η συμφωνία αυτή θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε περαιτέρω τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που κάνουμε. Και ε, καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταργήσει τους δασμούς για κάποια προϊόντα γεωργίας και αλλίες τα οποία βρίσκουν ήδη μια αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ε, είμαστε και οι δύο παραγωγοί ποιοτικών προϊόντων. 200 ευρωπαϊκά προϊόντα προστατεύονται στην Ιαπωνία και πάνω από 50 ιαπωνικά προϊόντα θα προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αριθμό αυτός θα αυξηθεί. Και η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί έτσι ώστε το σύστημα αυτό προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων να γίνει το ισχυρότερο από οποιονδήποτε άλλο εταίρων και βεβαίω το πεδίο συνεργασία στον τομέα τη γεωργίας για του παραγωγού μα είναι πολύ μεγάλο και καλωσορίζουμε το γεγονό αυτό. Και βεβαίω υπάρχει και το σχετικό κεφάλαιο στην συμφωνία αυτή. Για τα μη δασμολογικά μέτρα είναι γεγονό ότι οι δασμοί από μόνοι της δεν θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύ εξ αρχής ε, το επιζητούσε αυτό και η Ιαπωνία γνωρίζει την ε, σημασία του, αλλά οι πρακτικές αυτές ε, όμως δύσκολα βελτιώνονται. Ευτυχώς όμως καταφέραμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα στο να γίνουν τα συστήματα έγκρισης προδιαγραφών κτλ πιο διαφανή και προβλέψιμα σημαντικά ε, αποτελέσματα είχαμε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, των φαρμάκων, ε, των προσθέτων στα τρόφιμα και των χημικών προϊόντων. Και θα έλεγα πως μας βοήθησε αυτό, βοήθησε τις ρυθμιστικές αρχές να οδηγηθούν σε μια αμοιβαία κατανόηση. Κάτι το οποίο αποτελεί και μια καλή βάση για τη μελλοντική συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Οι δασμοί με την εξαίρεση λίγων, που έχουμε δει αυτή τη στιγμή καταργηθούν δεν επανέρχονται. Αλλά οι ρυθμιστικές διαφορές ε, είναι κάτι το διαφορετικό και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η υπόθεση. Οι οικονομικές δραστηριότητες αλλάζουν ε, και άρα οι κανόνες πρέπει να αλλάζουν. Πρέπει λοιπόν να συνομιλούμε συνεχώς για να εναρμονιστούν τα συστήματά μας και να γίνουν καλύτερα για την ε, μελλοντική αποτελεσματικότητά τους. Ήδη αναφέρθηκαν οι δημόσίε προμήθειε από τον κύριο Ντεμαρτή, δεν θα αναφερθώ. Και τέλος, επιλύσαμε το θέμα των σιδηροδρόμων. Ο κύριο Ντεμαρτή ανέφερε ότι ανοίξαμε τέσσερις άλλε πόλεις, 48 συνολικά, τώρα μιλάμε για 54 και θα ανεβεί ο αριθμός. είχαμε ανάλογες προσφορές και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε οι αγορές ε, των ε, δημοσίων προμηθειών ε, ανοίγουν. Τέλος, θα ήθελα να πω, όπως είπα και στην αρχή, ότι η πρόσβαση στην αγορά οπωσδήποτε ήταν σημαντική, αλλά τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον, που θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας και θα συνεχίσει αυτή να εμβαθύνεται, είναι πιο σημαντική το κεφάλαιο για την γεωργική συνεργασία, την ρυθμιστική συνεργασία είναι κάποια καλά παραδείγματα. Για τις επενδύσεις είχαμε πολύ σημαντικά εργαλεία, όπως αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Ντεμαρτή για την εταιρική διακυβέρνηση, που θα βελτιώσει το κλίμα και την θέση ε, δυνητικών επενδυτών που θέλουν να επενδύσουν και σε μικρές ε, και μεσαίες βιομηχανίες. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, να εμπαρόδω, πω οι άμεσε ξένε επενδύσει από την Ιαπωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει πάνω από μισό εκατομμύριο θέσει εργασία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ιαπωνία. Οπότε ε, έχουμε κάποιες δεσμεύσεις που έχουν γίνει πιο εύκολα κατανοητές όσον αφορά και τις επενδύσεις και τις υπηρεσίες. Οπότε οι δραστηριότητες αυτές καθιστούν την συμφωνία αυτή πιο σημαντική ε, σε σχέση με τα όσα επιτύχαμε στην πρόσβαση της αγοράς. Τέλος, δύο πράγματα ακόμα. Το ένα αφορά τις επενδύσεις. Υπάρχει μια ρήτρα για την απελευθέρωση των επενδύσεων που θα επιτρέψει στους δυνητικούς επενδυτές να αντιληφθούν πού βρίσκονται οι επενδυτικές ευκαιρίες. Όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, και το σύστημα αυτό επίλυσης διαφορών γνωρίζουμε τις ευαισθησίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Γι' αυτό αποφασίσαμε στο συγκεκριμένο αυτό θέμα να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με όλα τα σχετικά στοιχεία για να βγάλουμε τα καταλληλότερα συμπεράσματα στο μέλλον. Επίσης για την ροή των δεδομένων αντιλαμβανόμαστε όσον αφορά την ελεύθερη ροή δεδομένων και την σχετική προστασία της ιδιωτικότητας την σημασία του να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε την ρήτρα αναθεώρησης και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά το τι συμβαίνει στον ε, κόσμο για να προωθήσουμε την ιδιωτικότητα και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σουζούκη. Ε, τώρα έχουμε 20 λεπτά για ε, ρωτήσεις και απαντήσεις. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ στη θέση του κυρίου Βαλέσα που είναι ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Παρακαλώ κύριε Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, αλλά θα μιλήσω εξ ονόματος του Σκιώδους ε, Σεγγετού. Είναι μια τεράστια ευκαιρία λοιπόν, καταλαβαίνουμε και τις δύο πλευρές. Δεν θα επαναλάβω κάποια στοιχεία τα οποία ήδη έχουν υποθεί, αλλά θα εκφράσω μια πολιτική γνώμη όσον αφορά το μήνυμα ε, που ενέχεται αυτή τη μετατόπιση κατά του προστατευτισμού. Ε, και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση σήμερα στον κόσμο του εμπορίου. Άλλωστε το και ο κύριος ε, Σουζούκη λόγω ακριβώς της κυβέρνησης του Τραμπ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ιαπωνία μας υποστηρίζει στην απόφασή μας να παραμείνουμε αλληλέγγυοι και να ε, υπό τη σημαία του ελευθέρου εμπορίου. Και θα έχουν τη δυνατότητα τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ιαπωνία να προχωρήσουν γρήγορα στην επικύρωση της συμφωνίας. Και αναφερθήκατε στο ζήτημα των επενδύσεων. Θα ήθελα να ζητήσω μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το μέλλον ε, σε σχέση με την ε, διαπραγμάτευση της ε, συμφωνίας για τις επενδύσεις και πώς αξιολογείται το σύστημα το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι μελλοντικά μπορεί να είναι αποδεκτό από την Ιαπωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε και αναμένουμε με ανυπομονησία την επικύρωση της συμφωνίας. Αλλά έχω μια, ιδιαίτερη, μια δική ερώτηση για την ροή των δεδομένων. Και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η συμφωνία περιλαμβάνει μια σχετική ρήτρα προστασίας. Ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας θα συνεχίσουν εκτός του πλαισίου του FTA. Ε, το Μάιο οι επίτροποι είχαν μία συνάντηση στο Τόκιο. Ε, Ιδιομόλογοι, μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση σχέση με την ε, προστασία σπίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να αναφερθείτε στα ισχυρά σημεία αλλά και τις αδυναμίες αυτής της συμφωνίας ούτως ώστε να γίνουν κάποιες ε, βελτιώσεις όσον αφορά τη σύντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Ο Κλάους Μπούχνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα τρόφιμα. Η Ιαπωνία έχει πρόσθετα, πρόσθετες ουσίες ε, στα τρόφιμα που δεν είναι αποδεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι γιατί. Ε, και αυτό το ερώτημα δεν ε, περιλαμβάνει καμία αξιολόγηση. Απλώς θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά. Και αντίστροφα, τι γίνεται στην Ευρώπη έχουμε εμείς τα υψηλότερα, τις υψηλότερες τιμές όσον αφορά τη ραδιενέργεια ε, σχετικά με τη Φουκουσίμα και αν ναι, θα ήθελα να επισυνδύσω ότι ο Επίτροπος κύριος Έτιγκερ έδωσε κάποιες ε, προβλέψεις σε σχέση με τις οποίες θα υπάρξουν 900, 900 θάνατοι στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν κάποιοι θετική... Υπάρχουν κάποιες θετικές λίστες οι οποίες προτάθηκαν σε άλλα θέματα, για παράδειγμα στα χαρτιά, στα έγγραφα του Παναμά. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς κάτι σχετικό εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ. Ε, περιφέρειες όπως η δική μου στην ε, βορειοδυτική Αγγλία έχουν, σχετίζονται πολύ με την Ιαπωνία. Έχουμε 15 ιαπωνικές εταιρείε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά το Brexit βεβαίως και ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ε, συμφωνία με το Brexit. Η μεταβατική περίοδο θα είναι ένα θέμα ε, θα πρέπει να γίνει κάποια επαναδιαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε να προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο από τη συμφωνία αυτή. Ε, πώς, ε, από πού νομίζετε ότι θα μπορέσουν να προλάβουν αυτές οι βελτιώσεις. Είναι το καλύτερο δυνατό αυτό που έχουμε ή θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματικά να έχει κάποιους καλύτερους όρους. Το δεύτερο, όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο. Είπατε, κύριε Τομαρτή, ότι έχουν ενισχυθεί αυτές οι σχέσεις, αλλά όταν βλέπουμε το κείμενο έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με τη ΣΕΤΑ. Και όσον αφορά δε την εφαρμογή και την ρήτρα αναθεώρησης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κεφαλαίων σχετικά με το εμπόριο. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν ε, λιγότερες ε, προβλέψεις από ό,τι στη ΣΕΤΑ. Γιατί λοιπόν είπατε τότε ότι η συνθήκη αυτή είναι ισχυρότερη από τις άλλες. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη απευθύνεται προς τον κύριο Σουζούκη. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να αναφέρω ότι, ε, σημειώνω ότι δεν αναφερθήκατε στο θέμα των συμβάσεων του ΑΕΛΟ. Τώρα, η συμφωνία περιέχει μια δέσμευση για κύρωση των βασικών συμβάσεων ε, του ΑΕΛΟ. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε το τι γίνεται συγκεκριμένα στην Ιαπωνία για να πάμε προς αυτήν την κύρωση. Ξεκινώντας με αυτήν για την διακριτική μεταχείριση, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει και πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι η κύρωση αυτή θα συμβεί προσεχώς. Επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Ντεμαρτή. Είχαμε μία έντονη συζήτηση για την ΣΥΤΑ και παρά την συζήτηση βεβαίως είναι δύσκολο να βρούμε μια πιο προοδευτική εμπορική συμφωνία από αυτήν που υπογράψαμε με τον Καναδά, αλλά δεν τελειώνουν εκεί τα πράγματα. Το ερώτημά μου είναι ότι θεωρείτε ότι σε αυτήν την συμφωνία με την Ιαπωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να διατηρήσει κάποια υψηλά στοιχεία προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος θα λέγατε ότι είναι ένα βήμα προς τα εμπρός σε μια προοδευτική εμπορική ατζέντα. Ευχαριστώ κύριο Ντάκμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερωτήσεις έχω. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το επίπεδο και την αξία του εμπορίου που υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ιαπωνία. Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή θα αυξήσει το επίπεδο. Αν μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη. Τώρα, αν υπάρχει μια πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα, ε, πληρώνει η Ιαπωνία για την ενισχυμένη αυτή πρόσβαση. Η Βρετανική κυβέρνηση αναγκάζεται να πληρώσει, ενώ η Ιαπωνία όχι. Έχει κάποιες ουσιαστικές διατάξεις για τις υπηρεσίες η συμφωνία αυτή. Και τέλος, υπάρχει κάποια ρήτρα ελεύθερης ε, μετακίνησης ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Και επιπλέον η Ιαπωνία είναι κυρίαρχο κράτος που συμμετέχει στην παγκόσμια οικονομία αλλά έχει μια πολύ περιοριστική πολιτική για την ε, μετανάστευση. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να επιβάλλει τις αξίες της ε, στην ε, μεταναστευτική πολιτική της Ιαπωνίας. Και κάτι ακόμα. Έχω κάνει κάποιες πολύ λεπτομερείς τεχνικές ερωτήσεις και επί 8 εβδομάδες η Κομισιόν δεν απάντησε. Αν νομίζω το σύστημα λειτουργεί, εγώ δεν νομίζω ότι λειτουργεί, η Κομισιόν πρέπει να απαντά ε, στις ερωτήσεις ε, των Ευρωβουλευτών αντί να μην απαντά εντός των προθεσμιών που ορίζει το Κοινοβούλιο και εγώ. Ευχαριστώ Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά η εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία ήταν μια πλήρης εντολή, δηλαδή ε, περιλάμβανε τη Συμφωνία Επενδύσεων και στη συνέχεια αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι δύο συμφωνίες. Ποια είναι για σας η αποδεκτή προθεσμία για να καταλήξουμε σε μια Συμφωνία Επενδύσεων και ποια θα ήταν η μορφή που θα προσλάβει. Είναι πρόθυμη η Ιαπωνία να μπει σε μια πολύ τριμερή κούρσα επενδύσεων έτσι όπως την προβλέπει η Επιτροπή ε, είναι διατεθειμένη ε, λοιπόν η Ιαπωνία το κάνει και πότε. Δεύτερον, φαίνεται στο πλαίσιο των συμφωνιών απελευθέρωση των δασμών για τα προϊόντα της γεωργίας έχει μια μεταβατική περίοδο μέχρι 15 έτη. Ενώ η απελευθέρωση των προϊόντων που αφορούν ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή αυτοκίνητα της Ιαπωνίας ε, τα οποία εισάγονται προς την Ευρώπη είναι 7 έτη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά των μεταβατικών περιόδων μεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων Τρίτον, η, η Γερμανία είναι ε, ε, σημαντικός παίκτη εδώ. Γνωρίζετε τις αρνητικές και θετικές επιπτώσεις μιας μεγαλύτερης απελευθέρωσης σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πιο περιφερειακές. Και θέτω το ερώτημα προς τον κύριο Ντεμαρτή, όπως για παράδειγμα οι χώρες που έχουν υποφελθεί στο εσωτερικό της Ευρώπης από ορισμένες μετεγκαταστάσεις ε, βιομηχανικής παραγωγής, που ε, μπορεί να επηρεαστούν από έναν ανταγωνισμό ε, που να πρέπει από την Ιαπωνία. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον και τις κοινωνικές ε, προδιαγραφές, το να υπογραφεί μια συμφωνία του ILO που απαγορεύει την ε, καταναγκαστική εργασία θα έχει θετικέ επιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά ε, τα βάση και την προσπάθεια της ε, μη αποψήλωση των δασών, η Ιαπωνία εδώ δεν είναι πρόθυμη να συνεργαστεί. Ναι, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σούκη και όλους για την παρουσίασή τους εδώ. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω παρακαλώ. Πρώτον, όσο αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. τόσο ο κύριο Δεμαρτίο, όπω και ο κύριο Σούκη, ε, υπογράμμισαν πόσο σημασία έχει για τους μη δασμολογικούς φραγμούς αυτή η συμφωνία. Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση στην Ιαπωνική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να γνωρίζω πώς θα διασφαλιστεί ότι πράγματι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ιαπωνική αγορά και πώς θα λειτουργήσουν οι ισοτιμίες στην πιστοποίηση που επιτρέπουν ακριβώς ε, να έρθουν όλοι αυτοί οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Δεύτερη ερώτηση. Όλες οι εμπορικέ συμφωνίες προβλέπουν ή πρέπει να προβλέπουν μηχανισμούς που να τις βοηθούν να εξελίσσονται ανάλογα με τις συνθήκες κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει καθόλου μνήα για τη διάσταση του φύλου που θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες να υποφεληθούν από τη συμφωνία αυτή. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια βελτίωση στο μέλλον και με τι μηχανισμούς θα γινόταν αυτό. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο κύριος Γιάνφαλτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση αυτή, γιατί πραγματικά το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και χαίρομαι που τελικά η διαδικασία αυτή βαίνει προς την ολοκλήρωσή της. Ορισμένα ερωτήματα από την πλευρά μου τώρα. Το πρώτο ε, διατυπώθηκε ήδη από την κυρία Ρένα. Γι' αυτό δεν θα το επαναλάβω. Ωστόσο, ήθελα να τονίσω ότι και εγώ ενδιαφέρομαι πολύ για, την, ε, για το ζήτημα των επενδύσεων, το κομμάτι των επενδύσεων ε, της συμφωνίας. Και θα ήθελα να μας ενημερώσετε σε σχέση με την οπτική τόσο της Ιαπωνίας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επενδύσεις. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την πυρηνική ενέργεια. Η Ιαπωνία συνεχίζει να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την πηγή ενέργειας. Στην Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε, δίστανται απόψει τόσο όσον αφορά τη στρατηγική κατεύθυνση ορισμένων χωρών, για παράδειγμα η Γαλλία, η οποία χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια και άλλες χώρες όπως η Γερμανία που επιθυμούν μια έξοδο από την πυρηνική ενέργεια. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό έχει πολλά, είναι αμφίσιμο. Ε, στην Ιαπωνία το θέμα της πυρηνικής ενέργειας συνδέεται με κάποιες απειλές, ενδεχόμενες απειλές για τη χώρα και αυτό κάπως επισκιάζει τα πράγματα. Το τέταρτο ερώτημα αφορά ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, τόσο στην την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ε, χώρες του κόσμου. Τα, εργατικά, τα εργασιακά δικαιώματα. Ε, εδώ υπάρχουν ε, ριζικές διαφορές μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς. Θα δώσω το λόγο στο Ζαλίου και στον κύριο Σουσούκη για πέντε λεπτά παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο σε πέντε λεπτά να απαντήσει κανείς σε πάνω από δέκα λεπτά ερωτήσεις και μόνο, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις. Ναι. Οι διαπραγματεύσεις για την προστασία των επενδύσεων συνεχίζονται. Το λέω και στην κυρία Ρένα. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση κυρία Ρενά, δεν την ακούσαμε. Α, να σας απαντήσω γαλλικά. Ναι, ναι, θα ήταν πιο ευγενικό εκ μέρους μου, πράγματι. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζει στα γαλλικά ο ότι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το μείγμα, συνεχίζονται. Το σύστημα και το μείγμα είναι συνεπή μεταξύ τους αλλά διέπονται και από κάποια ανεξαρτησία. Ο στόχος του ΜΙΚ, δηλαδή του Δικαστηρίου του ε, Πολυμερούς για τις επενδύσεις, βάζει τις ίδιες προδιαγραφές για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών και χωρών σε πολυμερές πλαίσιο ακριβώς για να απλοποιηθεί το σύστημα και να μειωθεί το κόστος. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω εγώ ποιες είναι οι προθέσεις της Ιαπωνίας επ' αυτού. Πάντως, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία προστασίας επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ποτέ σε θέση να έχει συμφωνία προστασίας επενδύσεων που να μην περιλαμβάνει το σύστημα ICS και τις βασικές του αρχές. Αυτό είναι σαφές. Όσον αφορά τώρα, συνεχίζει στα αγγλικά ο τα άλλα στοιχεία, τις άλλες ερωτήσεις, σε ροή δεδομένων. Ναι. Υπάρχει αναθεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια νέα προσέγγιση για την ροή αυτή δεδομένων όπως γνωρίζετε. Η προσέγγιση αυτή δεν ήταν έτοιμη όταν ήμασταν σε διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και θα δούμε τώρα έγκαιρα κατά πόσο το στοιχείο αυτό θα περάσει από διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Αυτή η νέα προσέγγιση πάντως ε, κατετέθη για τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε τώρα με τη Χιλή και την Ινδονησία και η διαπραγματεύση για την καταλληλότητα των ε, δεδομένων συνεχίζεται στα πλαίσια των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Τώρα, κατά πόσο η συμφωνία αυτή προσθέτει ή αφαιρεί κάτι σε σχέση με τη συμφωνία ΣΥΤΑ. Κάθε συμφωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί ένα πλαίσιο, ένα πρότυπο και τώρα βασιζόμαστε στο σχέδιο των 15 σημείων που είναι απόλυτα συνεπές με ό,τι έχουμε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και για το DST με την Ιαπωνία υπάρχει κάτι θετικό σε σχέση με τη ΣΥΤΑ όσον αφορά το περιβάλλον, γιατί γίνεται μνήα της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη ΣΥΤΑ επί του παρόντος. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπει κάποια στιγμή. Και για την σύμβαση του, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας η θέση είναι γνωστή. Κανονικά είναι σαφές ότι το κεφάλαιο αυτό θα οδηγήσει και άλλη πλευρά να κυρώσει τις συμβάσεις του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Από εκεί και πέρα φυσικά οι Ιάπωνες συνάδελφοι πρέπει να απαντήσουν. Έρχομαι τώρα στην άλλη ερώτηση της κυρίας Αρένα για την μετάβαση. Υπάρχουν ε, διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με το προϊόν. Σε σπάνιες περιπτώσεις στη Γεωργία μπορεί να υπάρξει μεταβατική περίοδο μέχρι και 15 χρόνια. Συνήθως είναι μέχρι 10 χρόνια για τα ευαίσθητα προϊόντα, 7 χρόνια για τα αυτοκίνητα. Πρέπει να δούμε τη Γενική Συμφωνία, τη Γενική Ισορροπία της Συμφωνίας. Σήμερα 30% των εισαγωγών από την Ιαπωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χωρίς δρασμούς, ενώ είναι λιγότερο προς την άλλη κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό στην ισορροπία. Όταν πρόκειται τώρα για οικονομικές αναλύσεις, μια που αναφέρθηκαν άλλοι συνάδελφοι σε αυτό, το αποτέλεσμα δείχνει ότι η συμφωνία αυτή έχει ισορροπημένα αποτελέσματα και όσον αφορά τον όγκο του εμπορίου και όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει στο ΑΕΠ που σε απόλυτες τιμές είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Αυτά μπορώ να πω λοιπόν για τις οικονομικές επιπτώσεις. Εννοείται ότι είναι μια συμφωνία που όλες όλε συμφωνίες, που όπως όλες οι συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε, διέπεται από ισορροπία. Είναι ισορροπημένη συμφωνία. Όσον αφορά το θέμα της διάστασης του φύλου, υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, να έχουμε διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό στη συμφωνία με τη Χιλή θα δούμε κατά πόσο το πιλωτικό αυτό σχέδιο θα γίνει ο κανόνας. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσουμε από αυτή την πρώτη προσπάθεια. Νομίζω ότι έτσι έχω απαντήσει και έχω αφήσει και αρκετό χρόνο στο συνάδελφο. Ωραίο, κύριος Σουζούκη τώρα να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην καλύψω τις απαντήσεις που ήδη έδωσε ο κύριος Δημαρτή, αλλά όσον αφορά τις επενδύσεις, επειδή ρωτήσατε πολύ, η θέση μας όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων, κυρίως το στοιχείο που έχει να κάνει με τον μηχανισμό διευθέτησης διαφορών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να συμφωνήσει με στοιχεία ASTS. Οπότε πρέπει από εκεί, αυτό είναι το σημείο μας εκκίνησης, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε λογικά να βρούμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μελετούμε τα θετικά και τις αδυναμίες του ICS. Δεν λέμε ότι είμαστε εντελώ αντίθετοι, αλλά αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς πού είναι οι αδυναμίες αυτού του συστήματος. Να δούμε, μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανησυχίες. Για διμερείς συμφωνίες, το κόστος διατήρησης από μόνο του τέτοιων διμερών συμφωνιών είναι πολύ μεγάλο. Οπότε οι πολυμερείς συμφωνίες σαφώς και βοηθούν σε εξοικονόμηση κόστους. Αλλά θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα την ροή δεδομένων, Προσπαθούμε να δούμε τα συστήματά μας και πώς προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Όταν έχει ολοκληρωθεί αυτή η άσκηση θα μπορέσουμε και οι δύο πλευρές να αποφασίσουμε κατά πόσο μας καλύπτει η άλλη πλευρά και άρα έτσι να υπάρχει μια ήπια ροή δεδομένων. Πάντως συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που είναι δεσμευτικά. Ε, κάτι δεν άκουσα καλά γιατί πάλευα με τα ακουστικά μου ε, και το κουμπί. Κάτι ρωτήσατε για την πυρηνική ενέργεια, τη Φουκουσίμα. Μπορώ να σας πω πάντως ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Δηλαδή τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην Ιαπωνική αγορά έχουν επίπεδα ραδιενέργειας πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία είναι αποδεκτά στην διεθνή αγορά. Δεν μιλάμε βέβαια για προϊόντα τα οποία βρίσκονται παραπάνω. Το Brexit τώρα. Βεβαίως και είναι ένα σημαντικό ζήτημα για μας. Η βιομηχανική παρουσία της Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από πουθενά αλλού βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε φυσικά και μας ενδιαφέρουν οι διαπραγματεύσεις και θα θέλαμε να παραμείνει μια κατάσταση με ήπια σύνορα. Ελπίζουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν ήπια και κατά τη μεταβατική τουλάχιστον περίοδο να έχουμε κι εμείς ένα ρόλο και στο μεταξύ θα φροντίσουμε να διαπραγματευτούμε από μόνοι μας χωριστή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που ελπίζουμε να μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάπου συν, κάπου πλην. Πάντως θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στη Βρετανική αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο θέμα. για την Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 105-11 για τις διακρίσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πράγμα δεσμευτήκαμε στο κεφάλαιο που αναφέρεται στο εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη, εκεί που αναφέρεται δηλαδή η προστασία της εργασίας. Και στο εσωτερικό, αλλά όχι μόνο, θα ενισχύουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να εξετάσουμε περισσότερο σε βάθος την σχέση της εσωτερικής μας νομοθεσίας με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν δηλαδή από την κύρωση αυτής της συμφωνίας, της σύμβασης. Βέβαια προσπαθούμε να δούμε τι ισχύει κι αλλού και σε άλλες περιπτώσεις και θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Η, η Ιαπωνία όπως είπε και ο κύριος Δεμάρτη, ξέρω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που έχει δύο πλευρές. Ε, προφανώς και υπάρχουν ευαίσθητα προϊόντα. Έχουμε δεχτεί όμως, ε, έχουν γίνει δεκτές κάποιες δικές μας θέσεις για ευαίσθητα προϊόντα Έχουμε δεχτεί και έχουμε ε, λάβει και όλα την πρόσβαση των δικών μας ευαίσθητων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια προϊόντα τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε κάποια διέξοδο για τα προϊόντα, τα ευαίσθητα τα οποία παραμένουν σε συζήτηση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είτε πρόκειται για τις επενδύσεις, είτε πρόκειται για την πρόσβαση στην αγορά κλπ το ότι δεν αποτελούν μέρος του διεθνούς δικτύου, δεν έχουν πάντα τις πληροφορίες που θα έπρεπε, δεν ξέρουν πού να τις βρούνε. Αυτά είναι πράγματα που, με τα οποία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξέρουν πού μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η κυβέρνησή μας θα κάνει πάντως ό,τι μπορεί για να τις βοηθήσει. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα βέβαια από τη στιγμή που δεχόμαστε την σύμβαση όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία, συγγνώμη, του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για το ενεργειακό μας μείγμα για το 2030 ότι θα είναι τέτοιο που 20 με 22% θα βασιζόμαστε στα πυρηνικά και 20-24% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύουμε ότι η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική πηγή για την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Όπως διαπιστώσατε, αργεί πολύ το άνοιγμα ε, του πυρηνικού μας σταθμού, γιατί φυσικά θέλουμε να υπάρχει πλήρης ασφάλεια. Νομίζω ότι έτσι απάντησα, αλλά αν κάτι ξέχασα, συγγνώμη, προσπάθησα να καλύψω όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Σουζούκη. Ε, ελπίζω να έχετε περισσότερη τύχη με τους εταίρους σας στην Βρετανία γιατί μετά την παρέτηση χτες του Υπουργού Brexit μόλις μου ήρθε μήνυμα ότι παρετήθηκε και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Οπότε κανείς δεν ξέρει με ποιον ακριβώς θα συνομιλήσετε. Ναι, ναι, ο Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, ε, μόλις ξέχασα ότι όσον αφορά την ε, λαθροϊλοτομία μόλις ε, έχει εισαχθεί νομοθεσία που απαιτεί η παραγωγή προϊόντων ξυλίας να εγγραφούν και να αναφέρουν περιοδικά στο κάτος το ότι όσα αγοράζουν και πουλάνε προέρχονται από νόμιμη υλοτομία. Ναι, να το επιβεβαιώσω αυτό ότι οι διαδικασίες ε, για την υλοτομία ισχύουν επίσης και για το εμπόριο, αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ και στο στοιχείο γιατί μπορώ να δώσω την εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες τις ε, προφορικές και γραπτές ερωτήσεις. Για τις γραπτές ερωτήσεις θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο υπόθηκε τον κύριο Ντάρτμουθ. Ε, έχει απαντηθεί το ερώτημά σας πριν από μήνες. Υπάρχει στο site ε, από τις 15 Απριλίου και η άλλη σας ερώτηση απαντήθηκε το Μάιο. Οπότε, ε, δεν, δεν θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Θα ακούσουμε τώρα πέντε ειδικού. που θα μας ε, πούν κάποια βασικά πράγματα για την συμφωνία. Πέντε ειδικού όπως είπα. να τα δώσω πέντε λεπτά στον καθένα. Πρώτος είναι είναι η κυρία Λουίζα Σάντος, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της Business Europe. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Μια πολύ θετική συζήτηση σε μια ενδιαφέρουσα κάμπη για το εμπόριο και νομίζω ότι ίσως περνάμε σε μια νέα εποχή εμπορικών ε, σχέσεων οπότε ε, είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες του κλεισίματος ε, των αγορών και κάποιοι αποφασίζουν να επιβάλλουν δασμούς μονομερός αντί, για, αντί να συζητάνε και να συνεργάζονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες αγορές, νέες ευκαιρίες και πρέπει ακριβώ να βρεθούν νέε ευκαιρίε για τις ε, εταιρείε μας ε, μεγάλες και μικρές. Λοιπόν, θα τα κάνει αυτά αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι σήμερα μιλάμε για προσδοκίες, ε, Ποιε είναι οι δυνατότητες αυτής τη συμφωνίας, αλλά εξαρτάται από όλους μας να φροντίσουμε ότι πρώτα απ' όλα θα γνωρίζουν οι εταιρείε την συμφωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιαπωνία και ότι θα εκμεταλλευτούν αυτήν την συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να φροντίσουμε να γίνει γνωστή η συμφωνία και κατά την διάρκεια εφαρμογής της συμφωνίας να φροντίσουμε ώστε τα πιθανά ωφέλη αυτά να υπάρξουν στην πράξη. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας δώσω για τις ε, δυνατότητες και νομίζω το σημαντικότερο βήμα της συμφωνίας αυτής με την Ιαπωνία Βεβαίω ε, δεν είναι οι δασμοί. Οι δασμοί ήταν ήδη σχετικά χαμηλοί. Βεβαίω η Ιαπωνία πάντα παραπονιόταν για τα αυτοκίνητα. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε ψηλούς δασμούς στα καταναλωτικά αγαθά, ρούχα, παπούτσια και γεωργικά προϊόντα, οπότε νομίζω ότι θα υπάρξουν ωφέλη, αλλά το βασικό όφελος θα είναι σε τομείς όπως οι δημόσιες προμήθειες. Αναφέρατε την ρήτρα της επιχειρησιακής ασφάλειας, αλλά είναι ένας τομέας που όχι μόνο στις μεταφορές και τους σιδηροδρόμους, αλλά και σε άλλους τομείς θα δούμε ένα άνοιγμα της Ιαπωνικής αγοράς. Περισσότερες πόλεις θα ανοίξουν τις προμήθειές τους ε, σε ευρωπαϊκές θερίσματα Μετά για τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένας κέριος τομέας. Συνεργαζόμαστε με τους Ιαπωνές συναδέλφους μας και ακριβώς πρώτα απ' όλα σχεδιάσαμε τον αριθμό των μη δασμολογικών φραγμών. Εάν θυμάστε πριν ξεκινήσουμε είχαμε έναν μακροσκελή κατάλογο μη δασμολογικών φραγμών που ήταν όρος για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Ήταν λοιπόν σημαντικό ότι το είδε αυτό το ζήτημα η Ιαπωνία για να υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά ε, βεβαίω πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Δεν είναι θέμα επιλογών πολιτική. Ο καθένα θα μπορεί να συνεχίσει να κάνει τι επιλογέ του, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε λοιπόν σε βασικά ζητήματα, αυτοκίνητα, χημικά, ιατρικές συσκευές, ε, ψηφιακές συσκευές, θα πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο απελευθέρωσης της αγοράς που επιτεύχθη στις διαπραγματεύσεις και οι επιχειρήσει οπωσδήποτε θα παίξουν ρόλο και η κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα, οι καταναλωτέ ε, θα πρέπει να φροντίσουν κατά τη διάρκεια τη εφαρμογή να ε, διασφαλίσουμε ότι θα συμβεί αυτό. Ένα σημαντικό τομέα επίση όπου νομίζω ότι θα ωφεληθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αναφέρθηκε, είναι ο τομέα των υπηρεσιών. Και εδώ νομίζω, όταν μιλάμε για τους ανθρώπους ε, και αυτό όσον αφορά τις μεταθέσεις εντός των εταιριών και το ότι οι εταιρείες μεταθέτουν κόσμο. Ε, νομίζω ότι και εδώ πέρα παίζει σημαντικό ρόλο η συμφωνία αυτή. Ο άλλος τομέας ε, που είναι σημαντικός και αναφέρθηκε με το θέμα γεωργίας και τροφίμων δεν θα το αναφέρω αυτό γιατί θα το πούν οι συνάδελφοι αλλά το γεγονός ότι η Ιαπωνία αναγνώρισε πολλές σημαντικές γεωγραφικές ενδείξεις και εμείς αναγνωρίσαμε πολλές ιαπωνικές ανοίγει νέες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο το συγκεκριμένο δεν είναι διασφάλιση ότι θα ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά είναι σημαντικό Γιατί αν έχουμε ένα σημείο επαφή ε, και μια ιστοσελίδα για πληροφορίε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οπωσδήποτε βοηθάει. Και τέλο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Τώρα πρέπει να υλοποιηθεί και να φροντίσουμε κατά την υλοποίηση πραγματικά όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα για τις εταιρείες, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην Ιαπωνική πλευρά με τον κύριο Σιμίζου από την Κέινταν ε, Μεν, την Ιαπωνική Ένωση Επιχειρήσεων. Καλημέρα, ονομάζομαι Ακύρα Σιμίσου και είμαι πρόεδρος της Υποεπιτροπής για το Συντονισμό και τον Σχεδιασμό για την Ευρώπη. Ο κύριος Λάγκε, ε, κύριε Πέδρο Σίλβα Περέιρα και κύριε Μόνιμη Σιγητά για την Ιαπωνία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, κύριε Πιατκέτσεκ, και κύριε Γενική Διευθυντά της Γενικής Διεύθυνσης Trade και κύριε Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας για την Ιαπωνία και άλλα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να έρθω εδώ και να απευθυνθώ σε εσά για την σημασία που έχει η οικονομική αυτή εταιρική σχέση μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2007 το κέντ ήταν ε, ιδιαίτερα ενεργό όσον αφορά την σχέση των δύο πλευρών. Και γιατί, γιατί καταλαβαίναμε ότι η Ιαπωνία βρισκόταν πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα όμως ε, χαίρομαι που μπορώ να πω ότι με τη συμφωνία αυτή και χάρη στη σοφία των δύο πλευρών προχωράμε με ισορροπία, υψηλές προδιαγραφές και πρόοδο. Και είμαι πεπισμένο ότι αυτή η εμπορική συμφωνία θα βοηθήσει όχι μόνο να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά θα βοηθήσει να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και για τι δύο οικονομίες. Το δικό μας έθνος και οι εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κοινέ αξίε την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, την ε, ε, αγορά, την ε, ελεύθερη οικονομία και σεβόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κοινέ αξίες αυτές που αποτελούν και τη βάση εμπορικών συμφωνιών. Με κανόνες λοιπόν υψηλών προδιαγραφών για όλα, από το περιβάλλον και την προστασία ε, των εργασιακών δικαιωμάτων, την βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. Η συμφωνία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τόσο της Ιαπωνίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει και η προσδοκία ότι οι αξίες που υπογραμμίζουν ακριβώς αυτήν την ε, συμφωνία θα βοηθήσουν και στον θεμητό ανταγωνισμό και την πιο στενή ακόμα συνεργασία μεταξύ των οικονομιών των δύο χωρών, αλλά και των ε, ε, δύο χωρών αυτών και των αδειόμενων αγορών. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι 30% του παγκοσμίου και 40% του συνολικού εμπορίου είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όταν τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο παγκοσμιοποίηση, από τη μία και προστατευτισμού από την άλλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον που υπάρχουν τάσεις κατά τη παγκοσμιοποίηση και προστατευτισμός, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχουμε δηλαδή συμφωνίες με κανόνες που να διέπουν το διεθνέ εμπόριο. Χαιρόμαστε πολύ πάντως που έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ε, νομοθετική συνεργασία στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Από το 2012 και συνεργασία με την Business Europe, η Kay Darner, με τον εκπρόσωπο της Business Europe, την κυρία Σάντος, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις προκειμένου να προχωρήσουμε σε δραστηριότητες ρυθμιστικής, ε, ρυθμιστικού χαρακτήρα. Για να μειώσουμε τα μη δασμολογικά μέτρα, εναρμόνιση των ρυθμίσεων, των πρακτικών και πρόθεση αμοιβαίας αναγνώρισης προδιαγραφών και κανόνων σε τομείς όπως είναι τα φαρμακευτικά, τα ιατρικές συσκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Η βασική μας αρχή είναι να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς επιπλέον κόστος ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις επί του εμπορίου και των επενδύσεων. Συγχρόνως θέλουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της κάθε πλευράς να ρυθμίζει βάσει των δημοσίων πολιτικών σε τομείς όπως το, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ωφέλη του εμπορίου και ε, των επενδύσεων είναι υποφελή για όλους. Μια άλλη πλευρά της ρυθμιστικής συνεργασίας στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής είναι ότι προσφέρει την διαμόρφωση διεθνών κανόνων μέσα σε μια παγκόσμια οικονομική τάξη που είναι συμβατά με νέες τεχνολογίες και νέα πρότυπα επιχειρίζεστε. Ο δυναμικός ρόλος της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστιος και μπορούμε να θαρρύνουμε και να στηρίξουμε την έγκριση αυτής, ε, αυτών των κανόνων που διέπουν την εμπορική συμφωνία και στις υπόλοιπες οικονομίες. Και οι πρωτοβουλίες για αριθμιστική συνεργασία αποτελούν τη βάση ε, συζητήσεων με πολλές μεγάλες δυνάμεις που είναι γνωστές. Με δύο λόγια, η συμφωνία αυτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου οικονομικέ σχέσει Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέβουν σκαλοπάτι και προσβλέπουμε στην ε, υπογραφή, κύρωση και εφαρμογή τη συμφωνία αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο εμπειρογνώμων είναι ο κύριο Πεσόνεν, ο Γενικό Γραμματέα τη Κοπακατζέκα δηλαδή από την πλευρά, πράγματι από την πλευρά της ε, Γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να εκφράσω τις απόψεις των ε, Γεωργών όσον αφορά αυτή την ε, συμφωνία δεν μπορώ παρά να πω ότι συμφωνώ με, τους, ε, με το βασικό διαπραγματευτή της Ιαπωνίας όταν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία οδηγούν, ε, έχουν ένα ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη διατύπωση αυτού του πλαισίου συνεργασίας. Ενώ ε, και με, το, με την ευκαιρία αυτή θα υπάρξουν ε, και άλλοι εταίροι οι οποίοι θα προσχωρήσουν ε, σε αυτό το πλαίσιο. Ε, εμείς υποστηρίζουμε αυτή την περικτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας και είναι η συμφωνία με τις πιο, μαζικές, με τις πιο σημαντικές επιπτώσεις που έχει ποτέ υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα παράσχει τεράστιες ευκαιρίες για την εξαγωγή ε, τροφίμων ε, στην αγορά. Μαζί με τους Ευρωπαίους ε, εμπόρους θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή ενισχύει τον ρόλο των εταίρων μας και ε, βασίζεται σε μία απελευθέρωση του εμπορίου ε, σύμφωνα με κάποιους ε, κανόνες και προς και το, όφελος και των δύο πλευρών. Υπάρχουν κοινέ κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά την προσέγγιση του εμπορίου. Η οικογενειακή γεωργία στην Ιαπωνία είναι η βάση της παραγωγής και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή τροφίμων αλλά και στην ε, διαχείριση βασικών πόρων όπως είναι το νερό για παράδειγμα. Μαζί με τους Ιάπωνες συναδέλφους ε, δημιουργήσαμε την ε, Παγκόσμια Οργάνωση Αγρογεωργών και προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει με το ΠΟΕ. Οι Ευρωπαίοι και οι Ιάπωνες ε, καλλιεργητές συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίσουν όλες οι πολυμερείς ε, συμφωνίες να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της γεωργίας. Και βεβαίως σεβόμαστε πάρα πολύ τους Ιάπωνες συναδέλφους στο ρόλο τους. Ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, βεβαίως έχουν ένα σημαντικό ρόλο εδώ, είναι καθοριστικός παράγων, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ιαπωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσλάβει στρατηγικό ρόλο. Η εμπορική αυτή συμφωνία έχει υψηλό επίπεδο απαιτήσεων όσον αφορά την απομάκρυνση μη δασμολογικών φραγμών και πρόκειται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς όσον αφορά τρόφιμα ε, και ε, ποτά, για παράδειγμα, αλλά και άλλα προϊόντα. Ε, οι εξαγωγείς λοιπόν θα έχουν να αντλήσουν σημαντικά ωφέλη από αυτή τη συμφωνία. Ε, υπάρχουν βεβαίως κάποιες ευαισθησίες από την πλευρά της ε, Ιαπωνίας. Συνήθως ε, εξάγουμε προς την Ιαπωνία προϊόντα τα οποία δεν είναι ανταγωνιστικά με την εγχώρια παραγωγή. Για παράδειγμα, στον γαλακτοκομικό, στο γαλακτοκομικό τομέα. Ε, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θα μπορέσουν ε, να ασχολήσουν στην επονική αγορά εντελώς απαλλαγμένοι από δασμούς. Με 127 εκατομμύρια καταναλωτές, η Ιαπωνία είναι καθαρός εισαγωγές ορισμένων ευρωπαϊκών προϊόντων, για παράδειγμα τροφίμων. Ε, και υπάρχει και μία αυτάρκεια της 40%. Ε, είναι η, Ιαπωνία η Ιαπωνία η μεγαλύτερη αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που είναι μικρός προμηθευτής ε, γεωργικών ε, προϊόντων και έχει εισάγει η Ευρώπη μόνο 339 εκατομμύρια σε τέτοιες προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, τελευταία χρόνια διπλασιάστηκε αυτή η εισαγωγή και αφορά και εξειδικευμένα προϊόντα που είναι ενδιαφέροντα για την ευρωπαϊκή αγορά, όπως βόλιο κρέας υψηλής ε, ποιότητας. Ε, άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία διατύπωση υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, ε, θέματα υγιεινή, υγειονομικής ασφάλειας κλπ δεδομένου του υψηλού επίπεδου προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσπάθεια αυτή θα ωφελήσει και την Ιαπωνία και ενισχύουμε και τις δύο πλευρές να προσπαθήσουν για την αναγνώριση των διατάξεων του ΠΟΕ αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, κοινότητα των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ενθαρρυντικό και για τις ε, προσεχείς διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εξασφάλιση ισότιμων όρων εντό εντός της των Ευρωπαίων ε, παραγωγών. Επίσης χαιρετίζουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας για πάνω από 100, πάνω από 200, 200 γεωγραφικές ε, ενδείξεις ε, ε, όπως είναι για διάφορα για το ελλανδέζικο ουίσκι, για διάφορες μάρκες τυρί κλπ. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή επίσης προσδίδει μεγάλη σημασία σε θέματα περιφερειακού σε θέματα όλες τις περιφέρειες όσον αφορά ευρωπαϊκές συμφωνίες και θα είναι καλό παράδειγμα και για τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Είναι σημαντικό μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτή τη μετατόπιση και να επισπεύσει τη διαδικασία επικύρωσης σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για τους ε, γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να επισπευστεί η επικύρωση αυτής της συμφωνίας και είμαι πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή ε, θα παράσχει για την ευρωπαϊκή διατροφική αλυσίδα αξιόλογα αποτελέσματα αλλά και θα συνεισφέρει και στην ενίσχυση των χωρών των δύο πλευρών ε, δημιουργώντας αμεβαία ωφέλη ως ανταπόκριση στην αύξηση της ε, ζήτησης για προϊόντα υψηλής ε, ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πολύ και το γιαμασάκι ουίσκι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, προϊόν μεταξύ αυτών που αναφέρατε. τώρα από την Ιαπωνική Συνομοσπονδία ο κύριος Καβασίμα. Ναι. Αγγλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καβασίμα λέγομαι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, ε, κύριο τα μέλη του πάνελ, και για τα συλληπιτήριά σας για τις ε, καταστροφές που περνάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το Ρίγκο βεβαίω είναι το περιφερειακό κέντρο των συνδικάτων της Ιαπωνίας και προσπαθούμε ακριβώς να προστατεύσουμε τις ε, δουλειές ε, και το βιός όλων των εργαζομένων για να πάμε σε μια κοινωνία βιώσιμη και αναγνωρίζουμε την σημασία του να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος μας για να οδηγηθεί η Ιαπωνική οικονομία σε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία με απασχόληση. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προστατευτισμού στην διεθνή κοινότητα δεχόμαστε ότι, τα, ότι η σύναψη αυτής της ε, συμφωνίας ε, μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν το 30% του παγκοσμίου ΕΠ θα έχει μεγάλη σημασία για την προστασία του ελευθέρου εμπορίου και την πρόθεσή του. Και βεβαίως εμείς ε, ζητήσαμε οι προσπάθειες ε, της ε, κυβέρνησης να περιλάβουν και διαφάνειες διαπραγματεύσεις, να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις προδιαγραφές ασφαλείας μέσω κάποιων κοινών δηλώσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Οπότε υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο στην εμπορική αυτή συμφωνία για την βιώσιμη ανάπτυξη που έχει μεγάλη σημασία και και εμείς και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, ζητούν διαφάνεια και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στις ε, διαπραγματεύσεις και οι διοργανώσεις ανησυχούν ότι η τελική συμφωνία δεν περιέχει αποτελεσματικές διατάξεις ε, επιβολής των εργασιακών προβλέψεων και βεβαίως όσον αφορά τις 8 βασικές συμβάσεις του ΆΙΛΟ η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει δύο συμβάσει, την 105 για την καταναγκαστική εργασία και την 111 για τη διακριτική μεταχείριση. Και βεβαίως ζητάμε αυτό να διορθωθεί αμέσως και όλα τα μέρη ε, της Εμπορική συμφωνίας να σεβαστούν πλήρω και να εφαρμόσουν τις ε, διεθνεί συμβάσει για την εργασία. Η Ευρωπαϊκή και η Ιαπωνική Συνομοσπονδία Συνδικάτων θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ε, συμφωνία και να πιέζουν την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και την Ιαπωνική κυβέρνηση για να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτές είναι οι κοινέ δηλώσεις που κάνουμε. Οπότε στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα συνεισφέρει σε καλύτερη ποιότητα ζωής ε, για τους εργαζόμενους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και με την Ιαπωνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Λέα Άουφρετ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς είμαστε οργάνωση καταναλωτών με 43 οργανώσεις καταναλωτών σε 32 χώρες. Και συμμετέχουμε σε θέματα εμπορικά, γιατί τα εμπορικά θέματα και εμπορικές συμφωνίες έχουν επιπτώσεις στους καταναλωτές. Εννοείται. Καταρχήν, είμαστε υπέρ των συμφωνιών αυτών ελεύθερων συναλλαγών εφόσον έχουν απτά ωφέλη για τους καταναλωτές και υψηλά επίπεδα προστασίας. Τώρα η περίπτωση αυτή για τη συμφωνία με την Ιαπωνία τι προσφέρει στους καταναλωτές και σε επιχειρήσεις. Γιατί εμεί όταν καθορίζουμε τη θέση μας για ειδικέ εμπορικές συμφωνίες πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε στους καταναλωτές μας τι περιλαμβάνει. Για τη συμφωνία με την Ιαπωνία δυστυχώ δεν υπάρχουν πολλά ωφέλη για τον καταναλωτή. Εξού και είμαστε κάπω απογοτευμένοι και θα σα εξηγήσω γιατί σε λίγο. Τώρα με του ομολόγου μα στην Ιαπωνία, των συνδικάτων δηλαδή, καταλήγουμε σε ένα κατάλογο και τον δελάσουμε μεταξύ μας. Λέμε τι συμφωνίες θα ήταν εφικτές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Και όταν δούμε τα αποτελέσματα της συμφωνίας, δηλαδή με το δικό μας τον κατάλογο, βλέπουμε ότι παραμένουν πάρα πολλά ερωτηματικά, τελίτσες τελίτσες και κάποια σημεία και απογοητευτικά. Το πρώτο στοιχείο που θέλουμε εμείς στη συμφωνία είναι να δούμε πώς ε, θα τοποθετηθούν ακόμα καλύτεροι καταναλωτές στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Και παρόλο που υπάρχουν θετικά στοιχεία, ας πούμε για την ενημέρωση, για το roaming, ε, για την περιαγωγή δηλαδή, παρόλα αυτά όσα αναφέρονται είναι κάπως ασαφή και δεν υπάρχει καλός συντονισμός στα διάφορα κεφάλαια της συμφωνίας μεταξύ τους. Θα είχε νόημα σε εμπορικές συμφωνίες να έχει ο καταναλωτής μια συγκεκριμένη θέση. Να υπάρχει ένα κεφάλαιο για τους καταναλωτές, ας πούμε, όπως υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να υπάρχει και για τους καταναλωτές. Δεν λέω ότι το συστήνουμε για τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά σίγουρα για μια νέα. Έπειτα, θα έπρεπε να υπάρχουν απτά ωφέλη για τους καταναλωτές και προστασία είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ζητηθεί σε διάφορες γνωμοδοτήσεις. Από πλευρά τώρα του ωφέλους για τον καταναλωτή, θα πρέπει να δούμε τις τιμές των ιαπωνικών προϊόντων που θα έπρεπε να γίνουν πιο φτηνά. Όμως εδώ έχουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη ανάμεσα στην μείωση των δασμών και την μείωση της τιμής που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κοιτάζει, αλλά θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία εδώ. Γιατί δεν φτάνουν αυτά που έχουμε για να στηρίξουν οι καταναλωτές τη συμφωνία. Και τώρα έρχομαι στις κόκκινες γραμμές. Στις απαιτήσει μας. Εμείς θέλουμε η συμφωνία να προστατεύει τους καταναλωτές από την επίθεση ξένων επενδυτών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι διαχωρίζονται το εμπορικό σκέλος από εκείνο της προστασίας των επενδύσεων. Πάντως μια συμφωνία που να έχει ένα σύστημα δικαστηρίου για τις επενδύσεις που δεν επιτρέπει ε, σε κάποιον να προσφύγει επειδή πλήττονται οι κανόνες που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε να υπάρχει κάτι στο δημόσιο χώρο όπου να συμμετέχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα για τα τη ροή δεδομένων. Και εδώ έχουμε κόκκινες γραμμές. Θα έπρεπε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και χαιρόμαστε που γίνονται συζητήσεις για το πώς θα ήταν κατάλληλη η προστασία αυτή. Είναι ένα καλό πρωτοβήμα. Και υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης, αλλά θα έπρεπε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή. Αυτό είναι ένα άλλο ερωτηματικό μας. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια καλή προσέγγιση όσον αφορά τη ροή δεδομένων και την προστασία δεδομένων, χάρη βέβαια και στο καλό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά υπάρχει ερωτηματικό. Τι θα γίνει, πώς θα διατυπωθεί στη συμφωνία. Οπότε περιμένουμε πριν τοποθετηθούμε απόλυτα για τη συμφωνία. Συνοψίζω. Όσον αφορά το ωφέλη, δεν υπάρχουν σαφή ωφέλη για τους καταναλωτές δεν βλέπουμε πώς τοποθετείται καλύτερα ο καταναλωτής σε μια τέτοια συμφωνία. Δεν βλέπουμε βέβαια ούτε μεγάλες απειλές. Θα εξαρτηθεί πώς θα προχωρήσει η συζήτηση για τις επενδύσεις και τι θα γίνει με τη ροή δεδομένων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι είναι κρίμα που δεν μπορούμε ως οργάνωση καταναλωτών να στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε τα, οι καταναλωτές να ξέρετε ότι αλλού Ισλανδία, Αυστραλία έχουν κάπως καλύτερη θέση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πέντε λεπτά για ακριβείς ε, ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν προς τους εμπειρογνώμονες. Παρακαλώ. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη Ράγκο. Έχουμε επίγνωση των ε, προσπαθειών που κάνετε προκειμένου να έχετε την ε, επικύρωση της σύμβασης του ΆΕΛΟ. Ε, έχετε καθόλου ενδείξεις ότι κινούνται κάπως τα πράγματα, θα μπορούσε να συμβεί κάτι μελλοντικά, συγκεκριμένα όσον αφορά τη σύμβαση για τις διακρίσεις κατά των διακρίσεων. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία τους άλλους προσκεκλημένους μας. Ε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας και οι ανησυχίες σας όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η ρυθμιστική συνεργασία στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούχνερ έχει το λόγο. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, πρώτο ερώτημα όσον αφορά επίσης την ρυθμιστική συνεργασία είναι πράγματι το ορθό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν ε, τέτοιοι κίνδυνοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ο κίνδυνος όταν ε, ε, η νομοθεμησία μας είναι εξαρτημένη από ένα πλαίσιο όπου η οικονομία είναι ο καθοριστικός παράγων. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν εδώ να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καλά για τους πολίτες. Και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι υπονομεύεται η αρχή της ε, πρόληψης εδώ. Δεύτερο ερώτημα, τι γίνεται με τη ροή των δεδομένων μέχρι την ισχύ της ε, ρήτρας αναθεώρησης. Ε, θα ισχύσει έτσι όπως είναι στη συμφωνία, θα υπάρξουν περιορισμοί. Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων εν μέρη θα τεθεί εκτός ισχύω. Ωραία λοιπόν, τρεις βασικοί τομείς. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ίσως για τα εργασιακά δικαιώματα ο κύριος ε, Καβασίμα είναι ο αρμόδιος. Παρακαλώ κύριε Καβασίμα. Πιστεύω ότι η ερώτηση ήταν αν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ε, σχέση με το θέμα αυτό με την αντιμετώπιση της ε, σύμβασης. Γιατί η απάντηση δυστυχώ είναι όχι, γιατί η Ρέγκο ζήτησε από την Ιαπωνική κυβέρνηση να προβεί στην επικύρωση των ε, συμβάσεων αυτών. Βεβαίως ε, καταβάλουμε προσπάθειες ε, μαζί με την UTC και όπως είπε και ο κύριος Σουζούκη θα ήθελα να πω ότι είναι καλή ένδειξη η πίεση που ασκείται προς την Ιαπωνική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία, ποιος θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Όπως είπαμε στην αρχή, νομίζω ως επιχειρηματική κύκλη έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο, αλλά ήδη υπήρξε, υπάρχει μια προηγούμενη δομή εδώ, μια προηγούμενη οργάνωση. Μπορούμε να προτείνουμε κάποια πράγματα, βεβαίως σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπει η συμφωνία, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και άλλοι ενεχόμενοι εδώ, που είναι παρόντες εδώ, εισφέρουν και εκείνοι. Αλλά ως ε, επιχειρηματίε, επειδή γνωρίζουμε το κλάδο, γνωρίζουμε τι τεχνικέ πτυχέ. Είμαστε ε, διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με, τις, ε, ε, το, με, με τους διαφόρους κλάδους προκειμένου να φέρουμε τις σωστές προτάσεις στο τραπέζι. Επιτρέψατε μου να προσθέσω κάποια σχόλια. Είχαμε μια εσβάθος συζήτηση και βεβαίως αρχικά υπήρξαν κάποιες παρανοήσεις ε, και ε, ε, κάποιες αγωνιώτες προσπάθειες προστασία παλιάς αγορά, αγοράς. Αλλά τώρα υπάρχει μια αύξηση της αμοιβαίας αναγνώρισης και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής συμφωνίας θα περιβάλλουμε όχι μόνο τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα. Άρα λοιπόν το πλαίσιο αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή ε, μη αναμενόμενων κινδύνων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ρυθμιστική συνεργασία. Θα ήθελα να πω το εξή. Υπάρχει ένας ε, θετικός ε, διάλογος εκούσιος ε, μεταξύ των ρυθμιστών αλλά αυτό φορά το διάλογο εκτός της εμπορικής συμφωνίας. Ε, γιατί το πρόβλημα της ε, ε, το να επηρεάζει τη ρυθμιστική συνεργασία από την εμπορική συμφωνία είναι ο πρώτος στόχος να είναι η εμπορική απελευθέρωση και όχι η προστασία των καταναλωτών. Ε, βεβαίως γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν εκούσιο διάλογο, είναι θετικός ε, και έχουμε σημαντικές προσδοκίες. Ε και ε, ένα τέτοιο διάλογο θα υπάρξει και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και. Ε, ε, ο διάλογο αυτό μάλλον θα μοιάζει με αυτόν που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Τώρα. Έχουμε και το θέμα τη ροή των δεδομένων. Τι θα γίνει μέχρι να τέθει ενισχύ αυτό το κεφάλαιο. τρία χρόνια στο νέφο, τι θα γίνει. Είναι σαφής η διάταξη, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και αν ε, κανονικά υπάρχουν ροές δεδομένων ε, μεταξύ Ένωσης ε, και Ιαπωνίας θα συνεχίσουν όσο έχουν. Και θα υπενθυμίσω ότι το υπόδειγμα συμφωνίας που έχουμε τώρα και θα χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις μας αφορά πλήρη εφαρμογή της Γενικής Οδηγίας για την Προστασία των Δεδομένων. Δεν υπάρχει κάποια αμφισημία. Και κάτι άλλο. Υπάρχει πλήρης προστασία του δικαιώματος αυτού. Δεν μπορούν κάποιες εταιρείες να αμφισβητήσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και να υπενθυμίσω ότι ακόμα και στο παλιό SDS ε, που θεωρούσαμε κάπως ε, παροχημένο. Η Φίλιπ Μόρι έχασε από την Αυστραλία και την Ουρουγουάη και η Αυστραλία κέρδισε στον ΠΟΕ. Μάλιστα, οπότε σας ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η πρώτη έτσι, αρχή εξέτασης της συμφωνίας αυτής και θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα συνοψίσω εγώ την σημερινή συζήτηση. Αυτά θα τα αφήσω στο σχέδιο ψηφίσματος και συστάσεων που θα υποβάλω στο Κοινοβούλιο. Αλλά η ακρόαση επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Οι εντολές είναι δημόσιες, το κείμενο είναι γνωστό και θα γίνει έτσι μια σωστή συζήτηση και η προσοχή ε, ήταν σημαντική για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις οπότε τώρα απέχουμε έξι μήνες από την ε, τελική ψηφοφορία αρκετός χρόνος για να οριστικοποιηθεί το κείμενο και να ακούσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, η συμφωνία αυτή δεν είναι έκπληξη για το Κοινοβούλιο βεβαίως παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις εκφράζουμε τις ενισχύσεις μας αλλά και την στήριξη και βεβαίως θα πρέπει ακριβώ να δούμε ποιο είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω συναδέλφους ότι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στα τέλη Αυγούστου και βεβαίως ως μόνιμος συζητητής αναμένω και εγώ την συνεργασία με τους ε, συναδέλφους και τους κοιόδης συζητητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι θα έχουν τον χρόνο το καλοκαίρι στην παραλία να διαβάσουν την συμφωνία. Καλό να περάσετε λοιπόν. Έτσι ώστε τον Αύγουστο να ξεκινήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ειδικούς. Ευχαριστώ Ζαν Λούκ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σουζούκη που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ και καλή τύχη. So, ladies and gentlemen, please... Λοιπόν, κύριε και κύριοι, παρακαλώ, ησυχία. Δεν καταλαβαίνω γιατί φεύγετε από την αίθουσα. Αλλά θέλετε να φύγετε, παρακαλώ, ησύχω. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα 6. Ανταλλαγή απόψεων με την Χίλντε Χάρντεμαν, επικεφαλής των μέσων εξωτερικής πολιτικής για την διαδικασία Κίμπερλι. Χαιρόμαστε που είστε εδώ ε, μαζί μας. Είστε επικεφαλής ε, του μέσου εξωτερικής πολιτικής και θα μας πείτε για την πρόοδο που έχει σημειώσει η διαδικασία Κίμπερλι. Συγκεκριμένα ασκείται την Προεδρία ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Συνάδελφοι, θα θυμάστε ότι αυτό είναι ένα από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχουμε που μπορεί να επηρεάσει την βελτίωση της κατάστασης των διαμαντιών από περιοχές συγκρούσεων. Σημαντικό λοιπόν το θέμα. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για να σας πω λίγα πράγματα για τη διαδικασία αυτή ως πρόεδρος για το 2018. Η διαδικασία πιστοποίησης αυτή εισήχθη το 2003 για να σταματήσει η ροή διαμανδιών από περιοχές συγκρούσεων που πολλούνται για να χρηματοδοτήσουν συγκρούσεις. Σήμερα η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 54 μέρη και 18 κράτη. Πρόκειται για έναν εμπορικό κανονισμό της Ένωσης. Βασίζεται σε μια τριμερή δομή που περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα πέρα από τα κράτη. Είχε έναν θετικό αντίκτυπο. Το μερίδιο των διαμαντιών ε, στα κατέργαστα διαμάντια, των διαμαντιών συγκρούσεων, έχει πέσει από 15% το 2003 σε κάτω από 1%. Είναι κάτι το ουσιαστικό. Η διαδικασία αυτή επίσης βοήθησε να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να διαδοθεί η ιδέα ότι οι φυσικοί πόροι ανήκουν στις κοινότητες, ε, τις τοπικές και όχι στους ναι. ένοπλους ε, και βεβαίω υπάρχει και το πλαίσιο του ΟΣΑ με την δέουσα επιμέλεια. Ο αντίκτυπος λοιπόν αυτής της διαδικασίας μέχρι στιγμής ήταν ουσιαστικός αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια χαλάρωση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να παραμείνει ικανή να ανταποκριθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το 2011 κάναμε μια πρώτη προσπάθεια αναθεώρησης και προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάποιες κατευθυντηρίες γραμμές δεοντολογίας. Μια προσπάθεια η οποία δεν κατέληξε τότε. Το 2016 οι συμμετέχοντες άνοιξαν μια νέα διαδικασία αναθεώρησης που είναι ανοιχτή μέχρι το 2019. Οπότε το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την προεδρία της διαδικασίας και η μεταρρύθμιση είναι στο κέντρο της προεδρίας αυτής ως πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες εξυγχρονισμού της διαδικασίας αυτής και αποτελεσματικής μεταρρύθμισης η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τον Ιανουάριο να ασκεί την Προεδρία με δύο στόχους. Πρώτον, να υπάρχει μια συνοχή στην τριμερή δομή, δηλαδή κράτη επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών. Δεύτερον, να δώσει όθηση σε κάποιες πρωτοβουλίες για αύξηση της σταθερότητας ε, και της βιώσιμης ανάπτυξης ε, στις ε, εξορίξεις που στις μικρές κλίμακες εξορίξεις και τρίτον βεβαίω να προωθηθεί η σχετική ατζέντα έχουμε λοιπόν κάποια αποτελέσματα είμαστε στη μέση της διαδικασίας βεβαίω, η κοινωνία των πολιτών αναδιοργανώθηκε υπό την δυναμική ηγεσία της Αφρικής της Ζέλα, μια μήκυο από την Ζιμπάμπουη που έχει αναλάβει την ηγεσία της ε, κοινωνίας των πολιτών και θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Δεύτερον, οι χώρες ε, της λεγόμενης Ένωσης ε, του Ποταμού Μάνου, Λιβερία, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, σημειώνουν κάποια πρόοδο στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν καλύτερο διασυνοριακό έλεγχο και εφαρμογή του κράτους δικαίου στις ε, περιοχές όπου γίνεται η εξόριξη. Τέλος. Όσον αφορά τον οργανισμό που διαχειρίζεται την διαδικασία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέραμε σε μια αξιολόγηση αναγκών για να γίνει μια συζήτηση για μια μόνιμη γραμματεία και τέλος ως σύντονη μιας υπομάδας διαδικασία μεταρρύθμισης του βασικού εγγράφου, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει σημαντική πρόοδο στην καταγραφή οδηγιών και δηλώσεων και τεχνικών αποφάσεων. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι δομημένη και υπάρχει μία ενδιάμεση συνάντηση τον Ιούνιο και μία ολομέλεια το τέλος του έτους. Ε, έγινε λοιπόν η εξαμηνία συνάντηση στην Αμβέρσα και μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα και συγκεκριμένα να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση και τη μεταρρύθμιση. Η βασική προτεραιότητα είναι ακριβώς ε, το θέμα αυτό της μεταρρύθμισης ε, και Βεβαίω, περιλαμβάνεται εδώ και το πεδίο εφαρμογή τη διαδικασία αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να συνεχιστεί η δουλειά για την ανάπτυξη μια σαφού και πιστική προσέγγιση για την υπεύθυνη εξόρυξη διαμαντιών. Ο ορισμό των διαμαντιών από περιοχέ συγκρούσεων είναι πάρα πολύ βασικό για την πιστοποίηση και πηγαίνει χέρι με χέρι με την μεταρρύθμιση και τη ε, και τις σχετικές προκλήσεις. Όμως απαιτεί μια συνένεση και αντιλαμβάνεστε ότι 81 μέρη το καθιστούν αυτό δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επιτύχουμε κάποια πρόοδο και η θέση των εξορρυκτικών κοινοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη πρόσοχη στην συνεργασία, ειδικά όσον αφορά την εξόριξη σε ποταμούς και μικρής κλίμακας. Η αηφορία και η ευθύνη και η συμμετοχή στον διάλογο είναι σημεία αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως για να μπορέσουμε να λύσουμε διδάγματα από Έχουμε διδαχτεί στις διάφορες ε, κοινότητες. Ε, έχουμε και το σχετικό φόρουμ ακριβώς στο πλαίσιο της ευρύτερης διάσκεψης στην ε, Λουζάκα, στην Ζάμπια. Η Ολομέλεια του 2018 θα γίνει στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο από τις 12 μέχρι τις 16 μηνός. Η κυρία Μογκερίνη θα κηρύξει την έναρξη. Θα υπάρξει και ένα σχετικό φόρουμ και ακριβώς ε, θα είναι ένα φόρουμ το οποίο θα αφορά στατιστικά στοιχεία και ειδικού για την εξόρυξη διαμαντιών. Και όπως είπε και η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, η διαδικασία αυτή είναι ένα απόσπαστο μέρος της ε, δουλειάς μας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Για την ειρήνη, για να μην έχουμε νέες συγκρούσεις και να σταματήσει η χρηματοδότηση εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων και γεγονός είναι ότι θα πρέπει τα διαμάντια να παραγούν πλούτο και όχι σκλαβιά και είμαι στην διάθεσή σας ε, για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ωραία. Είναι μια άλλη πτυχή της εμπορικής πολιτικής και αυτή. Αυτά τα μέσα εξωτερικής πολιτικής βέβαια πρέπει να εφαρμόζονται. Ωραία, κύριε Χαουτάλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρτεμαν για τα όσα μα είπατε όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων τώρα που έχει την Προεδρία στη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αρχίσω με κάτι που δεν αναφέρατε και μετά θα σχολιάσω τα άλλα που αναφέρατε. Υπάρχει ένας κανονισμός του Συμβουλίου που δεν επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέκεται. Εντάξει, αυτό είναι θέμα εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά προβλέπεται αναθεώρηση όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να μην έχουμε απλώς ένα κανονισμό του Συμβουλίου, αλλά να έχουμε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα βοηθούσε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία, που είναι βασικό στοιχείο. Τώρα άκουσα διάφορα πολλά υποσχόμενα νέα από σας για το πώς προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, ώστε να αποτελέσει ένα στοιχείο και βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και ανθρώπων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά βέβαια, γιατί ακόμα και αν ο ορισμός της σύγκρουσης αναθεωρηθεί, δεν θα καλύπτει όλες τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είπατε τώρα ότι η άποψη της εξορρυκτικής κοινότητας είναι κεντρική σημασίας. Υπήρξε αντίσταση σε μια ευρύτερη κάλυψη που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Προεδρία της. Θα υπάρξει ρήτρα αναθεώρησης για τον κανονισμό Έπειτα, ο κανονισμός αυτός είναι 16 ετών ήδη με πολύ λίγες τροποποίησεις μέχρι τώρα. Οπότε το θέμα της δέωσας επιμέλειας πιστεύετε ότι φτάνει, ότι έχει υλοποιηθεί και ότι μας καλύπτει ή μήπως πρέπει να υπάρχουν περισσότερες υποχρεώσεις αναφορών εκθέσεων σε σχέση με την δέουσα επιμέλεια. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αναφερθήκατε στη Ζέλα από τη Ζιμπάμπουε. Όμως, μερικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ανυπόμονες με την διαδικασία και στον κανονισμό δεν υπάρχει τίποτα για το transit. Βάσει αυτού του κανονισμού αρχές μιας χώρας μπορούν να ελέγξουν ε, ε, φορτία transit για διαμάντια αν πιστεύουν ότι δεν συμμορφώνονται με τη διαδικασία Κίμπερλι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Ζήντσλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε όσον αφορά τη διαδικασία Kimberley. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία, να τη χρησιμοποιήσουμε καλά. Ε, δεν έχω όλα τα στοιχεία βέβαια και τα νούμερα για τη διαδικασία αυτή τα τελευταία χρόνια, αλλά εσείς είπατε ότι είχαμε πολλά και θετικά αποτελέσματα τελευταία, μετρήσιμα, γιατί εσείς έχετε στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να τα συνδυάσω όλα αυτά με το έργο εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ορυκτά σε ζώνες με συγκρούσεις. Ένα από τα συμπεράσματα στο οποίο εμείς εδώ καταλήξαμε είναι ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Άρα όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία, όπως συμβαίνει στη διαδικασία λέει τελικά. Είναι οι κυβερνήσεις, αλλά όχι μόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι επίσης οι δυνατότητες που έχουμε επιτόπου. Γιατί ό,τι και αν προσπαθούμε να χτίσουμε, όποιοι και αν είναι οι στόχοι της αναπτυξιακής μας πολιτικής, αν δεν έχετε ικανότητες επιτόπου, αν δεν έχετε εταίρους επιτόπου, δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό που θέλουμε τελικά στο κάτω-κάτω είναι ακριβώ αυτό, να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Και έτσι έρχομαι σε αυτήν την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογή τη διαδικασία Κίμπερλι, που ήταν πολύ περιορισμένο το 2002, αν δεν απατώμε. Είχαμε μια κατάσταση στην Αφρική και έπρεπε να συνεισφέρουμε να λυθεί. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, για παράδειγμα, θα πρέπει η διαδικασία του Κίμπερλεϊ να βοηθήσει τις χώρες εταίρους και περιφέρειες. Αναφερθήκατε στην αναθεώρηση και είπατε ότι είναι στους στόχους της διαδικασίας του Κιμπερλή. Μια τέτοια αναθεώρηση, μια τέτοια μεταρρύθμιση μπορεί να είναι εφικτή μόνο αν συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στο θέμα των διαμαντιών, όχι μόνο οι κυβερνήσεις. Η κατάσταση διαφέρει βέβαια από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες όπου δεν λειτουργούν οι κυβερνήσεις δεν μπορείς να τα λύσεις όλα στην πρωτεύουσα, ας πούμε, θα πρέπει να πας και στην περιφέρεια, να βρεις και άλλους φορείς και εταίρους εκεί. Και να συμπεριληφθεί φυσικά και η κοινωνία των πολιτών. Συνεπώς, αν κατάλαβα καλά, οι στόχοι της αναθεώρησης αυτής θα είναι πρώτα απ' όλα το πεδίο εφαρμογής, να διευρυνθεί, αν κατάλαβα καλά, και να εξυγχρονιστεί και η διακυβέρνηση της διαδικασίας Κίμπερλι. Πώς θα γίνει αυτό όμως. Είναι όπως και με τον ε, ΠΟΕ που βασίζεται στα μέλη. Όλες τις αποφάσεις την παίρνουν ομόφωνα τα μέλη. Δεν μπορεί να πάρει κανείς αλλιώς απόφαση με πλειοψηφία ας πούμε. Και άλλη μια ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προτάσεις για να υπάρξει μια μόνιμη γραμματεία της διαδικασίας Κίμπερλι που δεν υπάρχει προς το παρόν. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Υπάρχει πράγματι αυτή η δυνατότητα ή μόνο συζητήσεις γίνονται. Και αν υπάρχει θα πήγαινα πιο μακριά και θα ρώταγα είναι δυνατόν η μόνιμη αυτή γραμματεία να εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατασταθεί αυτή η μόνιμη γραμματεία. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Α, όχι, έχω και άλλες δύο. Έχω και άλλες δύο, λυπάμαι, αλλά έχουμε χρόνο, Πρόεδρε, έτσι. Λοιπόν, πρώτον, η διαδικασία Κίμπερλι συνεργάζεται με τον ΟΣΑ. Οπότε όταν μιλάμε για τη δέσου επιμέλεια και όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στις περιοχές με σύγκρουση σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η συνεργασία με τον ΩΣΑ. Ισχύει, βοηθάει και τέλος. Ίσως πιο δύσκολη ερώτηση, αλλά όλοι συζητάμε για την μετανάστευση αυτή την εποχή. Η μετανάστευση ήρθε για να μείνει. Είναι μια πρόκληση που θα παραμείνει. 5, 10, 15 χρόνια εδώ θα είναι. Όποτε εσείς πιστεύετε ότι κάποιες από αυτές τις χώρες είναι πηγή μετανάστευσης ε, οικονομικών μεταναστών έτσι, που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύετε ότι η διαδικασία του Κίμπερλι αν βοηθήσει να βελτιωθούν οι οικονομικές προοπτυχές των χωρών ε, αυτών που είναι πηγές μετανάστευσης θα βοηθούσε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές να έχουμε λιγότερη μετανάστευση λιγότερη μεταναστευτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις επόμενες δεκαετίες. Εντάξει, δεν λέω μεθαύριο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα απαντήσω τις ε, διάφορες ερωτήσεις από κοινού ε, θεματολογικά. Όπως αναφέρατε σωστά, κύριε Βίγκλερ, η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από ότι σήμερα όταν αντιμετωπίζαμε ολέθρους ε, πολέμους, εμφυλίους πολέμους, ε, ειδικά στη Δυτική Αφρική όπου τα διαμάντια χρηματοδοτούσαν ε, τους εμφυλίους πολέμους. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την, τη σχετική ταινία. Έτσι λοιπόν, αυτό το υπόβαθρο η διαδικασία Κίμπερλι συστάθηκε για να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, να μην πέσουν τα κατέρχαστα διαμάντια στα χέρια ανθρώπων ε, που χρηματοδοτούν εμφυλίους πολέμους. Και υπό την έννοια αυτή η διαδικασία Κίμπερλι υπήρξε πετυχημένη. Ε, και ήταν αποτελεσματική. Τώρα βρισκόμαστε 20 χρόνια μετά, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, την, να μετατρέψουμε τη διαδικασία αυτή και να την κάνουμε αποτελεσματική σε ένα διαφορετικό πλαίσιο τώρα. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της έσωσης επιμέλειας και το πώς η διαδικασία αυτή σχετίζεται με αυτό το οποίο συμβαίνει στον ΩΣΑ. Επίσης, το πώς ε, σχετίζεται με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ακατέργαστα διαμάντια που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Ε, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συνθετικών διαμαντιών που γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αγορά και υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι ε, ε, και υπάρχουν και σχετικές ανησυχίες στο ε, κλάδο της βιομηχανία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές αντιστάσεις και πολλοί δισταγμοί. Προκειμένου να αλλάξει η διαδικασία αυτή ε, και μέλη. Για πολλούς λόγους. Ορισμένοι φοβούνται ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι πλέον αποτελεσματική διαδικασία και θα εκπληρώνει το στόχο για τον οποίο έχει συσταθεί. Και βεβαίως ε, υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις όσον αφορά τη διεύρυνση του φάσματος προκειμένου να συμπεριληφθούν ανθρώπινα δικαιώματα ή εργασιακά ζητήματα στις χώρες παραγωγής αλλά ε, και στην Κίνα ή στην Ινδία που είναι σημαντική εταίροι στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και βεβαίω μπορείτε να κατανοήσετε ότι οι χρόνες αυτές είναι αρκετά απρόθυμες για αλλαγέ. Τώρα, όσον αφορά τη επιμέλεια στο πλαίσιο του ΙΣΑ, εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια προεθυμία να θεωρηθούν συμπληρωματικέ ε, διαδικασίες ε, ενώ η διαδικασία Κίμπελ θα ασχολείται με τα κατέργαστα διαμάντια και την προέλευσή τους και στη συνέχεια ο ΣΑ θα εξετάζει τα επόμενα βήματα στη διαδικασία και η βιομηχανία για πρώτη φορά ε, έλαβε μέρος στο παραδοσιακό Εαρινό φόρουμ του ΟΣΑ και είπε ότι θα ήθελε να συμμετέχει σε εκούσια βάση. Όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία Κέμπελη είναι οι κυβερνήσεις αυτές ε, που είναι οι βασικοί ε, συμμετέχοντες. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μια προσπάθεια συγχώνευσης, αλλά μια προσπάθεια αλληλοσυμπλήρωσης. Όπως είπατε, ε, πρόκειται εδώ για μια διαδικασία που βασίζεται σε, σε αρχή της ομοφωνίας. Έχουμε 83 ε, συμμετέχοντες, άρα οι αλλαγές εδώ δεν είναι πολύ εύκολες. Τώρα, όσον αφορά την ρύθμιση, ε, τον κανονισμό, συγγνώμη, τον κανονισμό που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρήσει τη διαδικασία Κίμπερλι σαν ένα βασικό τελωνιακό ε, κανονισμό. Υπάρχουν έξι περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κατέργαστα διαμάντια μπορούν να βγουν ή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το θέμα του transit ε, δεν είναι γύρι τόσα προβλήματα, γιατί εάν τα διαμάντια, ε, τα κατέργαστα μπουν μέσα στην Ευρώπη, θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτές τα, τις έξι περιοχές και το αντίστοιχο ισχύει και για τις ε, εξόδους των ε, διαμαντιών. Θα πρέπει να περάσουν από τα, τις έξι αυτές, ε, τις έξι, περιοχές. Άρα λοιπόν το θέμα του transit... δεν θεωρώ ότι εγείρει σημαντικά θέματα. Ο ίδιος ο κανονισμός δεν είναι κανονισμός, δεν είναι κανονισμός στην απόφαση. Ε, ε, βεβαίως ε, έχει μεγάλη αξία και θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμε προς την διαδικασία αναθεώρησης αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τον κανονισμό τους ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι ε, επιθυμητές ε, αλλαγές στο βασικό κείμενο. Αναφερθήκατε στο πεδίο εφαρμογής, ή ε, στο φάσμα μάλλον, στο πεδίο της διαδικασίας αυτές. Υπάρχουν πολλές χώρες παραγωγή, αλλά Εάν δούμε τον καταναλωτή, ε, διαπιστώνουμε ότι τα διαμάντια, ιδιαίτερα ως κοσμήματα, δεν είναι προϊόντα τα οποία αγοράζονται καθημερινά ε, και έχουν και εμείς ένα σημαντική φόρτιση. Άρα οι καταναλωτές ε, έχουν άποψη για την προέλευση των διαμαντιών που επιθυμούν να αγοράσουν και οι παραγωγές χώρες έχουν επίγνωση αυτής της κατάστασης. Αλλά προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο αυτό, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Και εφόσον θέτουμε το ερώτημα αν υπάρχουν αντιστάσεις, ναι, ε, απαντώ υπάρχουν αντιστάσεις από πολλές πλευρές. Ε, ανέφερα την Κίνα, θα μπορούσα να αναφέρω και τη Ρωσία, αλλά και χώρες παραγωγούς, όπως για παράδειγμα την Κεντρική Αφρική ή την Μποτσβάνα, ε, που έχουν ένα όνομα όσον αφορά την παραγωγή των διαμαντιών. Και η διαδικασία Κίμπερλι μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, λειτουργήσε σωστά, είχε αποτελέσματα και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου σε σχέση με τη σήμανση και λοιπά των προϊόντων, ε, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε στα θέματα αυτά. Και αν παρακεμίσαμε το πιάτο όπως είπε και ένας ε, βουλευτής εδώ, της διαδικασίας του Κέμπερλι, ίσως δεν θα είχαμε αποτελέσματα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια συζήτηση, να γεννήσουμε μια συζήτηση και να υπάρξει ένας προβληματισμός. Αλλά δεν βρισκόμαστε στο σημείο όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά τα διαμάντια. Και προκειμένου να είμαστε διαφανείς ε, προς όλους που επιθυμούν να συζητηθεί αυτό το ζήτημα, ε, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον ορισμό της περιοχής σύγκρουσης ε, υπό την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία Κίμπερλι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κατανοούμε ότι προκειμένου να δούμε, ότι θα πρέπει να ε, δούμε τι γίνεται με τις εξορεκτικές ε, κοινότητες. Ε, τα θέματα αυτά της χειροτεχνικής εξόριξης σε τέτοιες περιοχές είναι ένα ευαίσθητο θέμα και σχετίζεται και με την ζήτηση των ε, διαμαντιών. Βλέπουμε ότι, όπως σας είπα, ε, έρχονται στο προσκήνιο και τα συνθετικά διαμάντια, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται και συνεπώς αν γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία ε, ε, βλέπουμε ότι οι συνθήκες της εξορρυκτικής ε, διαδικασίας ε, βαίνουν στο περιθώριο και ανέρχονται άλλα ζητήματα στο θέμα της, της αγοράς αυτών των προϊόντων. Υπάρχει βεβαίως η επιθυμία από τις ε, παραγωγούς, από τις κοινότητες να τεθούν τα ζητήματα αυτά. Επίσης υπάρχει και η κοινωνία των ε, πολιτών, για παράδειγμα στη Ζιμπάμπε, ε, συγγνώμη, παίζει ένα σημαντικό ρόλο και υπάρχει αυτή η χειροτεχνική παραγωγή

εάν η διαδικασία αυτή θα, όταν συστάθηκε, είχε σαν στόχο να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση των εμφυλίων, τώρα αφορά περισσότερο την ε, κατάσταση των ηθαγενών ε, εξορρυκτικών κοινοτήτων. και τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει κάποιες διακηρύξεις οι έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας Κίμπελη προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των κοινοτήτων. Ε, ζητήσαμε, ε, υποβάλαμε μία ερώτηση προς την κυρία Χάουταλα εν σχέση με την εγκατάλειψη εκ μέρους ορισμένων ΜΚΟ των περιοχών αυτών. Για παράδειγμα, μια καναδική ΜΚΟ, η οποία ήταν επικεφαλής του συνασπισμού των ΜΚΟ, αυτοί έφυγαν λέγοντας ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα δουλεύοντας εκτός, όχι εντός των περιοχών αυτών. Και πιστεύουμε ότι είναι ε, και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ δραστήρια αφρικανική μικιό, η οποία προωθεί τα θέματα αυτά. Όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση και τη μόνιμη γραμματεία, θα ήθελα να απαντήσω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αλλά ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά ε, ταπεινοί ε, σε σχέση με την έδρα της γραμματείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Προεδρία της διαδικασίας του Κίμπερλι αλλά Μα ρωτήσετε κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρξει μια μόνιμη γραμματεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία ότι η έδρα θα πρέπει να είναι σε μια ουδέτερη χώρα. Και αν ε, δούμε ότι το 70% περνάνε ε, ε, από την Ευρώπη, από την Αμβέρσα συγκεκριμένα, ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τόσο ουδέτερη εδώ η Ευρώπη, όπως και η Βιέννη. Τώρα, όσον αφορά τις οικονομίες ε, των χωρών αυτών, όπου γίνεται αυτή η χειρονακτική εξόριξη, Ε, όπως σας είπα, ο ρόλος της μειώνεται. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει σημαντικά την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή τύχη εύχομαι στην διάσκεψη τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, διάλειμμα λίγων λεπτών για να σταματήσει η μετάδοση στο διαδίκτυο και να ακολουθήσει η συνεδρία σχετισμένη